Chers collègues, je propose de commencer notre... Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Πρώτο σημείο. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σας ενημερώνω ότι στην ψηφοφορία που, που θα έχουμε για το σημείο 18 και 23, που αύριο 9.30 θα ψηφίσουμε, πρέπει να εγκρίνουμε Επίσης για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών, ως ήθιστε, περιμένει τη δικιά μας γνωμοδότηση από αυτόν. Εξάλλου, θα εξετάσουμε ένα επιπλέον σημείο που είναι η κινητοποίηση του Ταμείου για τις κάτω χώρες. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα σχόλια επί της ημερησίας διατάξεως, θεωρείται εγκεκριμένη. Σημείο 2. Λέει Πρόεδρος, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής μας 25 και 26 Οκτωβρίου και 8 και 9 Νοεμβρίου. Αν δεν έχετε παρατηρήσει επ' αυτών μέχρι τη λήξη της συνεδριασιός μας, θεωρούνται και αυτά εγκεκριμένα. Τέλος, τις ανακοινώσεις της Προεδρού, σας ενημερώνω ότι η έκπληξη, ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Online. Αυτά με το πρώτο τμήμα της ημερήσιας διάταξης. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο 4. Περιμένουμε την Υπουργό, η οποία έρχεται από στιγμή σε στιγμή. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε. Όπως προβλέπετε, με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε εδώ την κυρία Ζέλε Μιλκέ, Υπουργό Απασχόλησης και Ισότητας. Θα μας παρουσιάσει τον απολογισμό της Βελγικής Προεδρίας, Γαλλικής είπε κατά λάθος η Πρόεδρος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια με την κυρία Όγκελινγκς θα έχουμε άτυπη συνάντηση 6 και 7 Δεκεμβρίου. Συμφωνήσαμε η συνάντηση αυτή να λάβει χώρα σε δύο στάδια. Πρώτον, θα συζητήσουμε τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η Βελγική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά θα ασχοληθούμε με το πακέτο Οικονομική Διακυβέρνηση, ΕΠΣΚΟ και ΕΚΟΦΗΝ. Κυρία Υπουργέ, σας δίνω το λόγο για το πρώτο αυτό τμήμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε ακριβώς για να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό, αν και είναι λίγο νωρί για απολογισμό, μια που έχουμε έναν ολόκληρο ακόμα μπροστά μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της Προεδρίας, ήδη έχουμε κάποια πράγματα πετύχει στα πλαίσια της Προεδρίας μας. Τον Ιούλιο ήμουν εδώ μετά πάλι από πρόσκλησή σας για να σας παρουσιάσω τους μεγάλους στόχους μας. Και τότε είπαμε ότι σε θέματα απασχόλησης οι στόχοι της Βελγικής Προεδρίας ήταν δύο ειδών. Είχαμε στόχους για την πολιτική απασχόληση, τους μεγάλους μας στόχους για την απασχόληση και στη συνέχεια κάτι άλλο θεμελιώδες και θα το δούμε στο δεύτερο τμήμα, στοιχεία οικονομικής διακυβέρνησης. Πώς δηλαδή θα φροντίσουμε να βάλουμε την απασχόληση και προτεραιότητα στις μακροοικονομικές μας ε, πολιτικές, αλλά πώς θα δούμε και την απασχόληση στα πλαίσια όλου αυτού του νέου μηχανισμού οικονομικής εποπτείας. Αυτό κάναμε. Είπαμε για την πολιτική απασχόλησης ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε δύο μεγάλες προκλήσεις, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, που αντιστοιχούν στις μεγάλες επαναστάσεις που ζούμε. Την πράσινη, η κλιματική επανάσταση, αν θέλετε, και την δημογραφική επανάσταση από την άλλη. Και γι' αυτό και αυτά τα δύο θέματα τα βάλαμε στην προτεραιότητα. Απασχόληση πράσινη και αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης που έχει να κάνει και με την απασχόληση, γιατί έχουμε πολλούς ε, μεγάλες ηλικίες ανθρώπους στην απασχόληση και θέλουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τις ανάγκες των υπηρεσιών μακροπρόθεσμα, δεδομένου ότι ζούμε περισσότερα χρόνια. Είπαμε επίσης τότε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε και στο θέμα της ισότητας στην απασχόληση. και ότι θέλουμε να δούμε και την προβληματική στα πλαίσια της εξωτερικής διάστασης της απασχόλησης. Μετά υπάρχουν και εγκάσια θέματα που έχουν να κάνουν με την αναδιάρθρωση και με τις μεταβάσεις, τις αλλαγές που θα δούμε σιγά σιγά μαζί. Ξεκινάω λοιπόν με το τι κάναμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Ποια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 και της οικονομικής διακυβέρνησης. Με αυτό βέβαια θα ασχοληθούμε πιο πολύ στο δεύτερο τμήμα της συζήτησης. Μετά θα κάνω τη σύνδεση με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που εγκρίναμε τον Οκτώβριο. Θα δούμε τι κάναμε με αυτά. Πράσινη οικονομία, πράσινες θέσεις απασχόλησης και δημογραφικές αλλαγές. Και τέλος, νομοθετικά, νομοθετικά ζητήματα που έχουμε νομοθετήσει δηλαδή. Την ε, Δευτέρα στο Συμβούλιο εξετάζονται διάφορα θέματα προς νομοθεσία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ποια είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και της οικονομικής διακυβέρνησης. Είναι περιττό νομίζω πόσο πολύ θεωρούμε και φαίνεται και από τα κείμενα ότι η απασχόληση πρέπει να είναι στην καρδιά της πολιτικής ανάπτυξης. Δεν πρόκειται μόνο για μια πολιτική ανάπτυξη, πρόκειται για μια πολιτική ανάπτυξη η οποία δημιουργεί απασχόληση. Και γι' αυτό και η λέξη απασχόληση βρίσκεται και στον τίτλο της στρατηγικής. Είτε πρόκειται για το 75% απασχόληση που θέλουμε να πετύχουμε το 2020, αλλά επίσης Πολλές κατευθυντήριες γραμμές συνδέονται άμεσα με τον στόχο αυτό. Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και όχι μόνο. Και στις οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές αναφέρεται. Για να μπορούμε να πετύχουμε λοιπόν αυτό το στόχο χρειάζεται μια οικονομική διακυβέρνηση η οποία να φροντίζει να είναι κατάλληλη και η πολιτική μας απασχόλησης. Στο άτυπο συμβούλιο του Ιουλίου, πολύ σημαντικό, ευαισθητοποίησαμε όλες τις χώρες μέλη για την προβληματική αυτή, δηλαδή η απασχόληση, πόσο μεγάλη σημασία έχει στα πλαίσια της νέας οικονομικής διακυβέρνησης. Τους δείξαμε βάσει κειμένου της Προεδρίας σε τι μεγάλο βαθμό οι πολιτικές απασχόλησης είναι ζωτική σημασίας μακροοικονομικά και ότι όλη, όλη αυτή η ανισορροπία που υπάρχει, διαβάζοντας ό,τι έχει γραφτεί όλα αυτά τα χρόνια δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει απασχόληση το να την αφήσουμε απ' έξω από την εποπτεία ή να την αναθέσουμε σε άλλους φορείς οι οποίοι δεν έχουν άμεση σχέση με την πολιτική απασχόληση θα ήταν λάθος. Ευαισθητοποίησαμε και τον Φαντορόν Πάο από αυτού. Μετά το άτυπο συμβούλιο ετοιμάσαμε ένα έγγραφο ως Προεδρία για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία τον Οκτώβριο εγκρίθηκαν στο συνέδριο Ευσκο για θέματα οικονομικής διακυβέρνησης, προκειμένου να έχουμε συστάσεις και πώς να εφαρμοστεί το 148 και να συμπεριληφθεί η απασχόληση στην οικονομική εποπτεία. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν περίμενα ότι θα τα καταφέρναμε, γιατί ήταν ένα επίμαχο θέμα. Καταφέραμε όμως να έχουμε συμπεράσματα που εγκρίθηκαν ομόφωνα στο Συμβούλιο μας για τις συστάσεις στην... σχετικά με την ε, οικονομική διακυβέρνηση. Να συμπεριληφθεί δηλαδή η απασχόληση και ομολογώ ότι με δυσκολία καταφέραμε να υπάρχει μνήμα στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου. Χρειάστηκε να αγωνιστούμε για καιρό για να πετύχουμε τη μνήμα αυτή. Υπάρχει πάντως. Και έχει μεγάλη σημασία. Θα συζητήσετε κι εσείς σύντομα για αυτό το θέμα και θα επανέλθουμε. Είναι λοιπόν η βασική προτεραιότητα αυτή της Βελγικής Προεδρίας. Θέλω τώρα να πω κάπως σε λεπτομέρειες για το τι κάναμε για την πολιτική απασχόληση και τις διάφορες πτυχές της. Κατευθυντήρες γραμμές πρώτα απ' όλα για την απασχόληση. Εγκρίθηκαν στις 21 Οκτωβρίου από το Συμβούλιο. Και είναι σημαντικό που δώσαμε αυτό το μήνυμα. Υπάρχει η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία δίνει νέο ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακόμα κι αν μερικές φορές είναι τυπικό, εμείς δεν το αντιμετωπίσαμε έτσι. Γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω από βάθος καρδίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον κύριο Ορή, την ε, πρόεδρο της Επιτροπής αυτής, για αυτά που καταφέραμε. Για το ότι περιορίστηκαν τελικά οι τροπολογίες στις πιο ουσιαστικές και εμείς ε, θελήσαμε να ενσωματωθούν στο βασικό κείμενο οι τροπολογίες αυτές που κρίναμε ότι ήταν καλές, κατάλληλες, ανταποκρίνονται σε μια πραγματικότητα και θεσμικά μιλώντας ήταν ένας νέος τρόπος να προχωρήσουμε η συνεργασία μας αυτή δηλαδή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τροποποίησαμε λοιπόν το κείμενο το οποίο τελικά εγκρίθηκε από το Συμβούλιο με όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, ε, παραγωγικότητα, συνοχή, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, αξιοπρεπείς ειδικές εργασίες, καταπολέμηση ενέργειας των νέων, ε, ένδια, μέρημνα για τα παιδιά κλπ. Εσείς βοηθήσατε πολύ, μας στηρίξατε και σε κάτι άλλο που είναι εθνική στόχη. Πολύ σημαντικό αυτό για μας και θα αναφερθώ αργότερα όταν μιλήσουμε για την μακροοικονομική ανάλυση. Υπάρχουν και οι πιο ευαίσθητες, πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συνδέονται όλα αυτά με την οικονομική διακυβέρνηση. Με την δικιά σας λοιπόν βοήθεια και στήριξη μπορέσαμε να τα συμπεριλάβουμε. Εγκρίθηκαν εν τέλει οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο θέμα που είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Οι σημερινές, δεν θα έλεγα οι αυριανές, που είναι αλλαγές στο κλίμα και δημογραφικές αλλαγές. Για το κλίμα πρώτα απ' όλα και την αγορά εργασίας. Προτεραιότητά μας ήταν βάσει του εξαίρετου έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στείλουμε ένα μήνυμα και να ζητήσουμε χτίσουμε μέτρα ή ένα πλαίσιο τέλος πάντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο χωρών μελών για την πράσινη απασχόληση. Αυτό ήταν ένα νέο θέμα. Θελήσαμε μάλιστα να το δώσουμε μεγάλη σημασία. Θα δείτε ότι οι δείκτες, τους οποίους θα αναφερθούμε όταν έρθουμε στη διακυβέρνηση, οι δείκτες αυτοί εγκρίθηκαν. Και βάσει Τη σωστή και καλή εργασία που έκανε η ομάδα εργασία ε, αναφέρεται το θέμα του πρασινίσματος των θέσεων απασχόλησης όλο και περισσότερο και στις διάφορες χώρες. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτή της δημιουργίας πράσινων θέσεων απασχόλησης βασιζόμενη και σε ποσοτικούς δείκτες αλλά και σε ποιοτικούς δείκτες. Βάσει λοιπόν των συστάσεων που αναφέρονται στην έκθεση Σρέντερ, Προχωρήσαμε στην διαπορκική μας διάσκεψη τέλη Σεπτεμβρίου για την πράσινη επασχόληση. Δύο μέρες πολύ ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές. Βάσει των όσων ακούσαμε, βάσει των στοιχείων που πήραμε από την Επιτροπή αλλά και από διάφορους διεθνείς οργανισμούς, καταλήξαμε σε συμπεράσματα. Είναι στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων της Δευτέρας. 6 Δεκεμβρίου, όπου η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη καλούνται να προωθήσουν την, ε, απόκτηση δεξιοτεχνιών, ενθαρρύνοντας ε, την ε, συνεχή κατάρτιση, τη διαβίω κατάρτιση. Περιλαμβάνουμε επίσης και την ιδέα του να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις να ξέρουμε τι θα ζητήσει η αγορά για να ετοιμάσουμε με τις κατάλληλες δεξιοτεχνίες τον κόσμο ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν στο μέλλον ώστε να μπορούμε να τις καλύψουμε και η πράσινη απασχόληση είναι βέβαια τέτοιου είδους ε, θέσεις απασχόλησης. Έχουμε την ιδέα να χρησιμοποιήσουμε τους δείχτες που σας είπα για να μετρήσουμε και για να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τα μέτρα που υιοθετούν τα κράτη-μέλη επ' αυτού. Στα συμπεράσματά μας επίσης τονίζουμε και το νέο ρόλο που έχουν οι υπηρεσίες απασχόλησης. Πώς πρέπει να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, πώς και τι ειδική προσέγγιση μπορούμε να έχουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς θα λάβουμε υπόψη μας και τα θέματα ασφάλειας στους χώρους εργασίας υγεία στους χώρους εργασίας. Γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας και την υγεία και ε, τα δύο φύλλα. Μερικές φορές ε, μέχρι τώρα συνηθίζαμε να λέμε ότι κάποιες δουλειές είναι πιο πολύ για τους άντρες. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε στο περιθώριο τις γυναίκες και να μην τους επιτρέπουμε να έχουν πρόσβαση στην πράσινη απασχόληση. Θέλουμε λοιπόν μέτρα ενθάρρυνσης προς τη σωστή κατεύθυνση που να έχουν να κάνουν και με τους μισθούς. Έπειτα, ε, φορολογική προσαρμογή, άμα θέλουμε να έχουμε μια οικονομία με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, πρέπει να φροντίσουμε να δώσουμε και φορολογικά κίνητρα αρκετά, ώστε να υπάρξει αυτή η πράσινη απασχόληση. Να λοιπόν, ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία θα παρουσιάσουμε στο Συμβούλιο τη Δευτέρα. Και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, μια πραγματική στρατηγική για το 2011, βάσει των διαφόρων συστάσεων. Η δεύτερη πρόκληση είναι η δημογραφική πρόκληση. Εδώ στα συμπεράσματά μας έχουμε συμπεριλάβει διάφορες προτεραιότητες. Το βασικό είναι η λογική Τη συμμετοχής των ε, πιο μεγάλων συλλογικών ανθρώπων στην αγορά. Και μην ξεχνάμε ότι αυξάνονται και οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται στους γυρότερους. Για το πρώτο, μιλάμε για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, για το ότι πρέπει να δουλεύουμε με καλές ηθικές εργασίας, γιατί και αυτό έχει μόνο στο τέλος της επαγγελματικής ζωής, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής. Δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις. Και πώς να επενδύσουμε στη διαβίου κατάρτιση, ώστε να προσαρμόσουμε την ε, κατάρτιση στις ανάγκες των ανθρώπων που είναι 45-50 χρονών και που δεν ακόμα στη σύνταξη. Θέλουμε να βελτιώσουμε δηλαδή την προσαρμογή μας και την ετοιμότητά μας στις αλλαγές. Κάναμε διάφορες διασκέψεις, στη Μαδρίτη για παράδειγμα για την απασχόληση και έχουμε και συστάσεις για να δώσουμε προτεραιότητα στην ποιότητα της απασχόλησης όταν πρόκειται για την φροντίδα, όταν πρόκειται για τις δουλειές στο νοσοκομείο, να φροντίσουμε για την ε, ε, για τις πιο πρόσκαιρες, την πιο πρόσκαιρη απασχόληση. Στις υπηρεσίες πρέπει να δούμε Επίσης, ποιες είναι οι νέες ανάγκες της υπηρεσίας. Και εδώ χρειάζεται διαβίου κατάρτιση και εδώ χρειάζεται η σωστή πολιτική κατάρτιση, ώστε να προσαρμοζόμαστε με προγράμματα δράσης ανακράτος μέλος και να βασιζόμαστε για αυτά σε ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ μας για να ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές. Τελικά, με την Προεδρία αυτή, τι έχουμε καταφέρει, που είναι και στην ημέρη διάταξη της 6ης Δεκεμβρίου, όπως σας είπα, για την ισότητα μισθών μεταξύ αντρών και γυναικών και για να μειωθούν οι διαφορές είναι κάτι που έχει να κάνει και με την απασχόληση και με την ισότητα. Εδώ λοιπόν έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. και από τη δουλειά της Επιτροπής, αλλά και για να προτείνουμε ότι πρέπει να περιλαμβάνει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να αναθεωρήσουμε όλους τους δείκτες που χρειάζεται. Και φροντίσαμε οι δείκτες αυτοί να επεκταθούν μάλιστα και περισσότερο βάσει της οικογενειακής κατάστασης. Πατρεμένος, ανήπαντρος, αριθμός παιδιών κτλ. Συστήνουμε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι αιτίε των διαφορών στους μισθούς και να βάλουν και μακροπρόθεσμους στόχους, ώστε από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους να πάψει να υπάρχει αυτή η διαφορά στους μισθούς μεταξύ αντρών και γυναικών. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν μια τέτοια, τέτοια μέτρα στις πολιτικές που θα υιοθετήσουν ε, μετά το Πάσχα. Έχουμε και κάποια συμπεράσματα αλλά αυτό ίσως σας αφορά λιγότερο, για την ισότητα ανδρών και γυναικών εκτός απασχόλησης και μισθών. Σε άλλους τομείς καταλήξαμε σε συμπεράσματα για την ποιότητα της απασχόλησης, για το λεγόμενο flex security, ευελιξία ασφάλεια. για την ποιότητα εργασία. Από κοινού με το Ίδρυμα του Δουβλίνου και με το Eurofonds ετοιμάσαμε αυτά τα συμπεράσματα και καταλήγουμε επίσης και σε συμπεράσματα σε θέματα θετικής μετάβασης Μιλάμε για τον φόρτο, τον σωματικό και τον ψυχικό που έχει να κάνει με την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Πώς να αισθάνεται κανείς καλά στη δουλειά του και πώς να συνδυάσει τον οικογενειακό με τον επαγγελματικό βίο. Αυτά είναι τα συμπεράσματά μας και νομίζω ότι είναι σημαντικά. Μερικές φορές τα αγνοούμε. Αυτά αγνοούμε αυτές τις πτυχές όταν μιλάμε για την απασχόληση. Εμείς στην κοινωνική διάσταση μάλλον την εξωτερική διάσταση, διορθώνει η κυρία Μιλκέ, τη θεωρούμε κάτι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για οικονομική διακυβέρνηση και για τη θέση της απασχόλησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχρόνως όμως πρέπει να κάνουμε το ίδιο και όταν μιλάμε για τη διεθνή διακυβέρνηση που έχει να κάνει με την μακροοικονομική πολιτική και εκεί πρέπει να ενισχυθεί η απασχόληση. Έχουμε λοιπόν σημαντικά συμπεράσματα που συνδυάζονται με τις συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Οργανώσαμε ένα φόρουμ με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για να ζητήσουμε να υπάρχει πιο συντονισμένη θέση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εκφράζεται έτσι στους G20, για παράδειγμα. Θέλουμε να ενισχυθεί ο ρόλος του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας όσον αφορά τις προδιαγραφές και τις συνθήκες εργασίας σε διεθνές επίπεδο. Συντάμε επίσης και ίσως η Γαλλική Προεδρία στο Τζίκοση μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Πρέπει συστηματικά να έχουμε συνεδρίαση των Υπουργών Απασχόλησης πριν από τα G20. Γιατί, για να εξηγούμε κάθε φορά γιατί η απασχόληση πρέπει να είναι στην καρδιά του G20. Θέλουμε να στηρίξουμε και τις εταιρικέ σχέσεις και το περιφερειακό επίπεδο. Παρά τις πολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, καταφέραμε παρόλα αυτά να έχουμε τους υπουργούς απασχόλησης στα πλαίσια της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης, όπου ζητήσαμε την ενίσχυση της εταιρική σχέσης και για την απασχόληση. Διότι έτσι μπορούμε να έχουμε κοινέ ευαισθησίε και να υποστηρίξουμε από κοινού διάφορε ιδέε και σε διεθνέ επίπεδο αλλά και σε επίπεδο G20. Να λοιπόν, που έχουμε φτάσει. 13 και 14 Δεκεμβρίου θα έχουμε και το ΖΕΜ και εκεί θα συζητήσουμε για την εξωτερική διάσταση. Αυτά όσον αφορά το δεύτερο τμήμα, λοιπόν, που έχει να κάνει με τις προτεραιότητές μας έτσι όπως τις καθορίσαμε για την απασχόληση. Και θα ολοκληρώσω με το νομοθετικό μας έργο. Εδώ δεν έχω να σας πω πολλά, δυστυχώς, αλλά είναι δύσκολο να προχωρήσουν ε, μερικά πράγματα, παρόλο που πολύ θα ήθελα να είχαμε πάει πιο μακριά. Έχουμε να κάνουμε με την οδηγία και τα δικαιώματα των ε, λεχόνων. Θέλαμε να αλλάξουμε την αρχική πρόταση, να πάμε στις 20 εβδομάδες για την άδεια μητρότητας, ε, με πληρωμένη άδεια και να μιλάμε και για γονική άδεια. Και επίσης στην οδηγία αυτή θέλαμε να περιλαμβάνεται και η ιδέα της ε, άδειας του πατέρα. Νομίζω ότι είναι απόλυτα θεμητή αυτή η στόχη. Τα κράτη-μέλη δυσκολεύονται. Επειδή βέβαια το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι αυτό που είναι, το γνωστό. Τα ελλείμματα, η λιτότητα. Υπάρχει μεγάλος φόβος ότι τα κράτη δεν θα μπορέσουν να αναλάβουν το κόστος μιας τέτοιας οδηγίας. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε, πρέπει να φροντίσουμε η συζήτηση αυτή να καταλήξει με έγκριση της πρότασης. Μπορεί να μην έχει οριμάσει ο χρόνος, το καταλαβαίνουμε. Θελήσαμε όμως να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Οργανώσαμε τη Δευτέρα στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ συζήτηση με συγκεκριμένα θέματα για να κάνουμε προτάσεις ως Προεδρείο και να δώσουμε ιδέες για κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων μπορεί να προχωρήσει η συζήτηση υπό Ουγγρικής Προεδρίας και σίγουρα επί Πολωνικής Προεδρίας. Και έτσι το 2011 να καταλήξουμε σε πρόταση αφού έχει προηγηθεί διάλογος με το Κοινοβούλιο εννοείται. Η ιδέα λοιπόν είναι, η ιδέα, λοιπόν, είναι η συζήτηση αυτή να οδηγήσει σε κάποια κεκτημένα. Προοδευτικά μπορούμε να προχωρήσουμε στον χρόνο, αλλά ίσως μπορούμε να πιέσουμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ έχω συζητήσει και με την κυρία Στρέλα για το δημοσιονομικό ζήτημα. Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους, αλλά βλέποντας πότε μπορούμε να βάλουμε στόχους για μετά το 2020 ή για πριν το 2020 και να προχωρήσουμε σιγά σιγά εφαρμόζοντας την οδηγία ε, ίσως σε τρία-τέσσερα χρόνια. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις ή αναλλακτικές προτάσεις για τις επόμενες προεδρίες. Όσον αφορά την οδηγία για την ισότητα, πιστεύω ότι αφορά λιγότερο την Επιτροπή σας. Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικά προβλήματα που μπλοκάρουν τα πράγματα, αλλά θέλουμε μία έκθεση τουλάχιστον για την διάκριση όσον αφορά την κατοικία, τις διακρίσεις ε, στην κατοικία και για τις δημοσιονομικές υπηρεσίες. Εδώ μπορούμε να προσφέρουμε κάποια, νομίζω, επιτεύγματα για την μετανάστευση, την οικονομική μετανάστευση, που δεν είναι βέβαια άμεσα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλησα να παρουσιάσω κάτι για το πόσο έχουν προχωρήσει τρεις προτάσεις οδηγίες όσον αφορά την οικονομική μετανάστευση που βρίσκονται στο Υπουργείο Πασχόλησης επί του παρόντος για την ICT και τους εποχιακούς ε, ε, εργάτες. Υπάρχει τεχνική ομάδα για την μετανάστευση που ασχολείται με αυτά και πρόκειται να έχουμε μια δεύτερη συνεδρίαση μέσα Δεκεμβρίου. Θέλουμε για το σημείο αυτό η Ουγγρική Προεδρία να το ολοκληρώσει. Αυτά για το πρώτο τμήμα που είχα να σας πω, πλην δηλαδή της οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα που προσπαθήσαμε να προωθήσουμε υποβελικής Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε και για την συνενοχή που δημιουργήσατε με αυτό το Κοινοβούλιο και με αυτή την Επιτροπή, έτσι ώστε προ, για πρώτη φορά να μπορέσουμε να έχουμε κατευθυντήρε γραμμές για την απασχόληση που να αντικατοπτρίζουν την ποιότητα της συζήτηση ε, που θεσπίσαμε και νομίζω ότι από την πλευρά του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου είναι ένα σημαντικό στάδιο. Θα το ξανασυζητήσουμε για να δούμε πώς αυτή, βάσει αυτής της πρώτης επιτυχίας θα μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα. Είπατε πόση σημασία προσδίδεται στην εξωτερική διάσταση και εγώ θέλω να σας πω ότι σε αυτή την Επιτροπή, όπως τα γνωρίζετε, έχουμε μία έκθεση υποεκπόνηση ο κύριος Φάλπ είναι ο αρμόδιος συζητητής. Και θα έχουμε κατά νου ε, φωνή της ε, Υπουργού Υποθέσεων και Απασχόλησης και Ισότητας να λαμβάνεται υπόψη ε, και στις διαπραγματεύσεις ε, στο ΠΟΕ και στη δική μας συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις. Νομίζω ότι η ιδέα είναι να έχουμε μία συνεδρίαση υπουργών απασχόλησης όπως ήδη έγινε πριν από τη συνεδρίαση G20. Είναι κάτι που το υποστηρίζει αυτή η Επιτροπή. Ιδίω αν ε, δούμε τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα αυτής της πρώτης εμπειρίας. Είναι αρκετά ενδιαφέροντα και έτσι θα σταλεί μια αντιπροσωπεία της δικής μας επιτροπής ε, στη Νέα Υόρκη κατά την ε, ημερίδα που οργανώνεται για την εξάλληψη της φτώχειας. Καθώς αυτό το θέμα μας απασχολεί. Έχω ήδη ένα μακρύ κατάλογο ε, βουλευτών που έχουν ζητήσει το λόγο να δώσω το λόγο δύο στους συναδέλφους και κατόπιν θα επανέλθει το κύριο Τόμας Μαν και κατόπιν ο κύριος Σέρκας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Προεδρία του Συμβουλίου ε, των ε, φίλων μας των Βέλγων είχε να περάσει και από τις συμπληγάδες όλες αυτές τις ε, προσπάθειες συγκρότησης κυβέρνησης. Τώρα έχω μια ερώτηση. Γιατί είναι τόσο δύσκολο για τις χώρες μέλη να ασχοληθούν με τις ποσοστώσεις. Είπατε κι εσείς ότι για τους δείκτες μπορούμε να συζητήσουμε. Μπορούν να περιληφθούν οι δείκτες. Και οι χώρες μέλη φαίνεται διατεθειμένες να <clears throat> τους δεχθούν. Γιατί όμως για τις ποσοστώσεις δυσκολεύονται τόσο πολύ. Έχουν την εντύπωση οι χώρες μέλη ότι θέλει να αναμειχθεί η Ευρώπη υπερβολικά γιατί είναι σωστό ότι χρειαζόμαστε ορισμένες ποσοστώσεις για τα όσα θέλουμε να επιτύχουμε. Εγώ είμαι σαφώς υπέρ της αρχής της επικουρικότητας, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό επίσης να φροντίσουμε να πούμε ότι πρέπει να επιτύχουμε κάποιο κοινό περιθώριο. Αν το επιτύχουμε αυτό θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Τώρα, μέσα στο έτος 2010, αγώνας κατά της φτώχειας, ένα από τα item είναι η μείωση του αριθμού, του ποσοστού δηλαδή των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Αυτό, σα το θυμίζω, ήταν ένας κοινό στόχος. Δεύτερο, ποια είναι η αξία των εκθέσεων ιδία πρωτοβουλία και δίπλα μου εδώ η κυρία Σρόιντερ έχει κάνει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για τις λεγόμενες πράσινε θέσει εργασία που βρήκε μεγάλη απήχηση μέσα στο Κοινοβούλιο και έχουμε κάνει και άλλες για να υπάρξει μια δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών. Τι θέση έχουν αυτές στην ε, εργασία του Συμβουλίου Υπουργών. Θεωρούν ότι απλώς είναι, θέση, είναι εκθέσεις του Κοινοβουλίου, δηλαδή δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένα ψήφισμά του, ή τις λαμβάνουν ω βάση για κάποια παραπέρα δουλειά. Απλώς δηλαδή τις λαμβάνουν υποσημείωση και μετά δεν ασχολούνται περισσότερο οι υπουργοί. Ο κ. Σέρκας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συντομία. Ε, θα ήθελα να πω ότι και εγώ θέλω να εκφράσω την ε, ε, ευχαριστή μου για την παρουσία της ε, Υπουργού εδώ και μπορώ να πω ότι η δική μου εμπειρία είναι ότι πολύ ικανοποιημένο από την πολύ μεγάλη προσοχή που μας έδωσε η Βελγική Προεδρία αλλά και για την προσπάθεια που κάνετε για να προχωρήσουν πολύ δύσκολοι φάκελοι. Εσείς μιλήσατε για την πολιτική απασχόληση, για την απάντηση που θα δοθεί στα δημογραφικά προβλήματα της Ευρώπης και για τα πιο καυτά θέματα του. Ε, ε, νομοθετικής ε, πρωτοβουλίας. Ε, βρισκόμαστε φυσικά σε μια οικονομική κρίση και ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη έχουν μονή για τα επίγοντα θέματα και διακινδυνεύουμε να αφήσουμε σε δεύτερο πλάνο σημαντικά θέματα και αυτά τα θέματα τέθηκαν στην ημερήσια διάταξη χάρη στις δράσεις της Βελγικής Προεδρίας και θέλω να το τονίσω εγώ σήμερα εσείς δεσμευτήκατε και ακούσατε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβούλιο ενώ το Συμβούλιο είχε ακολουθήσει μία άλλη επικίνδυνη οδό να διατηρεί σε ε, όλα αυτά τα γεγονότα μία διακυβερνητική θέση και να μην αναγνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης ε, με το Συμβούλιο σε αυτή την ε, νέα διάσταση της Ευρώπης των πολιτών. Μιλάμε για μια Ευρώπη όχι μόνο των κρατών αλλά και των πολιτών και παρά τις προσπαθίες ε, δυστυχώς ε, πάντοτε ε, βλέπουμε ότι στο Συμβούλιο δεν λαμβάνονται συστηματικά τα επιχειρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε καν μας απαντούν. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια από τα σημαντικά θέματα που προωθήσατε, όπως είναι η εννέα άδεια για τα μεταναστευτικά. Αυτό το θέμα σημείωσε σημαντική πρόοδο χάρη στις προσπάθειες που έκανε η Βελγική Προεδρία αλλά και που θα συνεχίσει να κάνει υπό το τρίο, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο και μπορούμε να έχουμε μια πολύ μεγάλη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αρκεί το Συμβούλιο να καταλάβει ότι όταν έρχεται η στιγμή να νομοθετήσουμε για θέματα που αφορούν ε, ουσιαστικά δικαιώματα των ατομών, δεν μπορούν να υπάρχουν παρεκκλήσεις τα οποία δεν δικαιολογούνται ε, στην κοινωνία των πολιτών, ε, στους πολίτες, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ε, δεν ε, ε, μπορούμε εδώ πάντοτε να εμφανίζουμε ένα επιχείρημα ή το παρνήσι του το και πάντοτε πρέπει να ξαναγκάζεται να υποχωρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί το Συμβούλιο ποτέ δεν δέχεται καμία από τις δικές μας προτάσεις. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Μιλκέ Ταμάλα και ελπίζω τους επόμενους μήνες να συνεχίσουμε να έχουμε τη δική σας συνεισφορά για να ολοκληρωθούν κάποια από τα θέματα τα οποία θα θέλαμε θέλαμε να δούμε να έχουν ολοκληρωθεί τώρα, αλλά δυστυχώ θα περάσουν στι επόμενε προεδρίε. Α ακούσουμε ακόμη ένα μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Όλοι έχουν εγγραφεί ούτω ή άλλω. Κύριε Σέντερ Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Βελγική Προεδρία για την παρουσία της εδώ. Ευχαριστώ πολύ και για την καλή συνεργασία. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν αξιέπαινος ο τρόπος με τον οποίο εργαστήκατε μαζί μας, ειδικά στον τομέα της πράσινης εργασίας, του δημογραφικού, σε δύσκολα θέματα, σε δύσκολα τοσχέ. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι επίσης για ορισμένα θέματα διακρίσεων. Γνωρίζουμε ότι ορισμένες χώρες μέλη έχουν στυλώσει τα πόδια για λόγους ιδεολογικούς, αλλά μπορούμε να βγούμε και να πούμε και στους ψηφοφόρους μας ότι πραγματικά περάσαμε μια βελική προεδρία η οποία κατέβαλε σοβαρές προσπάθειες. Χαίρομαι κιόλα που σχετικά με τις πρωτοβουλίες που εγκρίναμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις λάβατε σοβαρά υπόψη σας. Κάτι που δεν συμβαίνει πάντα, γι' αυτό λοιπόν εκφράζω ιδιαίτερη ικανοποίηση. Και μάλιστα αυτό βγήκε ως μήνυμα και προς τα έξω. Θα ήθελα ωστόσο να ρωτήσω κατά πόσο η δική σας δέσμευση στα θέματα αυτά που είναι τόσο σημαντικά την συμμερίζονται και οι άλλες χώρες μέλη. Ή μένουν μοναχά στα χαρτιά ότι θα τα εφαρμόσετε στο Βέλγιο είμαι πεπισμένη διότι σας είδα τόσο στρατευμένη ε, για τα θέματα αυτά στην εθνική σας πολιτική που γι' αυτό είμαι πεπισμένη. Αλλά υπάρχει κάποιο ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών μελών που να βγουν και να πούνε Όχι, εμεί είμαστε οι καλύτεροι, εμεί θα τα εφαρμόσουμε καλύτερα τα πράγματα αυτά στην εθνική μα πολιτική. Και ε, πώς θεωρείτε ότι πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται το Κοινοβούλιο για να προωθήσει παραπέρα αυτές τις πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Μάν. Ναι, πιστεύω ότι η ερμηνεία σας για το φόβο των κρατών μελών ε, είναι πραγματική. Υπάρχει ένας φόβος παρεμβατισμού στις εθνικές πολιτικές, ε, ενώ αν ε, το δούμε από τη σκοπιά της αποτελεσματικότητας, αν χρησιμοποιήσουμε σωστά την έννοια των στόχων με τους ανεξάρτητους και αποτελεσματικούς δείκτες, νομίζω ότι όλοι θα είμαστε κερδισμένοι. Εγώ πάντοτε υπεράσπιζα την ιδέα να έχουμε ε, στόχους αριθμητικούς και υποστόχους, όμως νομίζω ότι υπάρχει ένας φόβος, κυρίως όταν μιλάμε για κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης Δηλαδή και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εμπόδιο και θα φτάσουμε και στο δεύτερο τμήμα ε, της παρουσίασης μου. Αυτό έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση. Νομίζω ότι συνδέονται τα δύο ζητήματα, ενισχύονται οι φόβοι από το συμπληρωματικό βάρος που μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της οικονομικής αποπτίας σε ό,τι αφορά τώρα τη των ε, πράσινων θέσεων εργασία και τις δημογραφικές προκλήσεις να σας πω ότι στα συμπεράσματά μας ε, κάνουμε μία και στο δικό σας ψήφισμα που μας ενέπνευσε τα μάλα. Επίσης, να απαντήσω και στην κυρία Σρέντερ Οπότε δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα συμπεράσματα. Εμεί δεν θέλουμε να έχουμε ε, φιλολογικού χαρακτήρα συμπεράσματα. Θέλαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι, γιατί πρέπει να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση για να ζητήσουμε καταρχήν από την Κομισιόν να αναλάβει δράση βάσει των δικών σα ψηφισμάτων, που ήταν ιδιαίτερα ρεαλιστικά, μα επηρέασαν ε, και εμεί περιμέναμε και πολλά από την Κομισιόν μάλιστα για να παρουσιάσει μια στρατηγική για τι πράσινε θέσει εργασία. Αλλά ε, και αυτό είναι το σημαντικό της συζήτηση που κάνουμε προηγουμένως. Ε, ίσως ε, ο καλύτερος τρόπος να μπορέσουμε να έχουμε μόνιμα αυτές τις προοπτικές είναι να τις εγγραψούμε μέσα στους δείκτες και στο scoreboard. Και ε, ελπίζουμε αυτά να αποτελέσουν ε, σημαντικά εργαλεία για τη διακυβέρνηση αύριο. Αυτό στα εργαλεία που εθετούμε εμεί είτε μιλάμε ε, για εργαλεία της Επιτροπής Απασχόλησης, γιατί απαιτήθηκε να υπάρχει μία στις πράσινες θέσεις εργασίας και Επίσης, ε, παράλληλα έχουμε και το Ευρωπαϊκό Ξάμεινο και την ε, σχετική οικονομική εποπτεία και ε, στα πλαίσια των κατευθυντηρών γραμμών έχουμε όχι μόνο τους δείκτες για τις πράσινες επεσχόλες που θα χρησιμοποιηθούν από την ΕΜΚΟ συστηματικά αύριο, δηλαδή θα έχουμε μια συστηματική ανάλυση των προτεραιοτήτων, έτσι θα καταδείξουμε ότι υπάρχει προσέγγιση για τις πράσινες εργασίες και υπάρχει ανάλυση ανάλυση. Έτσι λοιπόν ε, θα δούμε και θα συγκρίνουμε πώς προχωρούν ε, τα κράτη-μέλη και τι προτάσεις έχει κάνει η Κομισιόν και σε ό,τι αφορά την ε, γύρανση για τους διάφορους δείκτες που πολύ γρήγορα και επαγγελματικά προετοιμάστηκαν από την ΕΜΚΟ. Έχουμε το προφίλ δικτών για έναν αριθμό εργαζομένων από τα 50 έτη για να δούμε τις εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα από την ηλικία αυτή. Τώρα, όσο όσα είπε ο κύριο Σέρκα, ε, ναι, αλήθεια είναι, έχουμε μία εξέλιξη νοητική, έχουμε και τη συνθήκη, αλλά έχουμε και τις πολιτικές εξελίξεις στη σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και γι' αυτό στην ε, παρουσίαση που θα κάνω για να εισαγάγω τη συζήτηση για την οδηγία για τη μητρότητα. Θα πω ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ε, τι λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο εκπροσωπεί τόσα εκατομμύρια πολίτες και ε, νομίζω ότι ε, ε, τώρα, γιατί δεν έχουμε τα μέσα, δεν μπορούμε να παγώσουμε τη λήψη της απόφασης. Κοιτάξτε, μπορούμε να την τροποποιήσουμε, να την καταστήσουμε πιο συμβατή και με το δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε και θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα λογική εταιρική σχέση με το Κοινοβούλιο, τουλάχιστον αυτό διαπίστωσε η Βελγική Προεδρία, γιατί ήταν και η πρώτη Προεδρία υπό κανονικό καθεστώς. Ε, δηλαδή είχαμε διατρέξει ένα πλήρες εξάμεινο από τη Σύνθεση της και είδαμε πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτό το θέμα των δεσμεύσεων όπως αναφερθήκαμε και στην ενιαία άδεια, στις πράσινες και κτλ. Αυτό δεν θα έλθει από τις ε, υπουργικές ομάδες ε, του Βελγίου, αλλά πρόκειται για δεσμεύσεις ε, οι οποίες θα συνεχίσουν να προωθούνται καθολικά. Μας μένουν 40 λεπτά και ακόμη 6 άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι για να έχουμε και το χρόνο να μπούμε και στο δεύτερο θέμα της συνάντησης μας. Κύριε Γκρουμ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πώς σκοπεύετε να δώσετε περισσότερη προβολή σε αυτό το ταμείο, όπως ανακοίνωσε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σε ό,τι αφορά τώρα την απασχόληση των πιο ηλικιωμένων. Ε, τι έχετε σκεφτεί για την ε, υγεία και την ε, ασφάλεια στο χώρο εργασίας, γιατί φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλος αντίκτυπος αυτών των θεμάτων και τρίτον για την μητρότητα και την άδεια μητρότητας. Μην ανησυχείτε, σε λίγο θα φύγω. Τώρα για την άδεια μητρότητα, εμείς θέλαμε 18 εβδομάδες με μερική πληρωμή, όμως ε, ε, εσείς ανακοινώσατε ότι θέλετε να προσφέρετε βοήθεια στις γυναίκες ε, σε ό,τι αφορά τον τρόπο φύλαξη των παιδιών και την περίοδο και σε σχέση με την υιοθεσία, ε, δηλαδή να έχουμε ισότιμο, ισοδύναμο καθεστώς με την άδεια μητρότητα. Κύριε Όρη και κατόπιν κυρία Ελίνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας κύριε Υπουργέ για την παρέμβασή σας. Θυμούμε στις αρχές της Βελικής Προεδρίας ότι θυμούμε πως αρχίσαμε και ε, τελικά πόσο καλά συνεργαστήκαμε με πόσες προτάσεις του Κοινοβουλίου ε, δεχθήκατε. Ελπίζω η επόμενη Προεδρία να προσεγγίσει τα θέματα αυτά με τον ίδιο επικοδομητικό τρόπο. Ε, τα θέματα που αναπτύξατε κυρία Υπουργέ είναι σημαντικά. Θα ήθελα να γνωρίζω ε, επειδή μάλιστα ακόμα δεν έχουμε δει τα διάφορα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, ποια από αυτά δηλαδή υλοποιήθηκαν πια ίσως όχι, αν υπήρχε δηλαδή συνένεση και στο Συμβούλιο αλλά και εδώ, νομίζω ότι η Βελγική Προεδρία πάντως έχει αρχίσει την εκπόνηση των πρώτων σχεδίων για τη μεταρρύθμιση. Θέλω να μάθω τι ε, θεωρείτε, για, τι, τι γνώμη έχετε για την λεγόμενη flex security, για την κατάρτιση των άνω των, μετεκπαίδευση μάλλον των άνω των 50 ετών Νομίζω σε διάφορα ε, όργανα που ασχολούνται με την απασχόληση και που συναντώνται συχνά. Είναι σωστό αυτό, σωστή η τάση αυτή και είναι θετικό επίσης να ανατίθενται μελέτες για την καλύτερη εξέταση των θεμάτων αυτών. Η Ουγγρική Προεδρία επίσης αναμένει τα πορίσματα των μελετών αυτών και η ερώτησή μου επίσης είναι τι προπαρασκευαστικές ενέργειες κάνετε σε συνεργασία με την Ουγγρική Προεδρία για να συνεχιστούν, να συνεχιστεί η πορεία αυτή και να επιτεθούν και άλλα βήματα στην επόμενη Προεδρία. Α, Λίν, ευχαριστώ, ευχαριστώ ε, και εσάς κύριε Υπουργέ για την συνεργασία μαζί μας. Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου για να μείνει η ε, οδηγία για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και τις επιρροές τους εκτός. Βέβαια, τώρα ε, επίσης για την ε, μητρική, για την μητρική άδεια, πολλοί ψήφισαν στο Κοινοβούλιο υπέρ των 20 εβδομάδων με πλήρη αμοιβή. Βέβαια κατανοώ ότι λόγω της οικονομικής κρίσης κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί και δεν ήταν και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στην ε, πλειοψηφία. Μιλήσατε τώρα για τις ε, διακρίσεις και για τα ισότιμα δικαιώματα. Έχουμε πλησιάσει σε μια ε, έγκριση από το Συμβούλιο. Να σταματήσουν δηλαδή να εμποδίζουν την πρόοδο ορισμένες χώρες μέλη. Ευχαριστώ για την ε, πολύ ευρία εισαγωγή στα θέματα που κάνατε, λέει η κυρία Τούρουνεν. Μια συγκεκριμένη ερώτηση σε σχέση με την ανεργία των νέων, που είναι ένα από τα θέματα των τριών προεδριών Ισπανικής, Βελγικής και Ουγγρικής. Ε, στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, νεολαία εν κινήσει, μέσα στο 2020 δηλαδή, ζητεί από το Συμβουλίο να δώσει εγγυήσεις για την απασχόληση των νέων. Που θα λέει δηλαδή ότι οι νέοι δεν ε, μπορούν να μείνουν στην ανεργία παραπάνω από τέσσερις μήνες και θα πρέπει να έχουν ε, εγγυημένη θέση σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή σε απασχόληση. Αυτό είναι κρίσιμο για τους νέους. Ρωτώ λοιπόν, υπάρχει η δυνατότητα είτε εσείς είτε οι Ούγγροι να υποβάλουν την σύσταση αυτή του Συμβουλίου όπως έχει ζητήσει η δική μας Επιτροπή, όπως έχει ζητήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τους νέους όλης της Ευρώπης. Κύριε Λενικεβιτσιούτε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει κυρία Μπλίνικεβιτσιούτε. Σας ευχαριστώ και σας κύριε Υπουργέ για την παρουσίαση και την ανάπτυξη των θεμάτων επί των οποίων εργαστήκατε. Πιστεύω και εγώ ότι ήταν καλή η συνεργασία μας, κυρίως για την ανεργία. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που λάβατε υπόψη πολλές συστάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι όλες βέβαια. Εφιστώ την προσοχή σας στο εξής. Ως Προεδρία, ίσως θα έπρεπε να δώσετε περισσότερη προσοχή στους ηλικιωμένους και στην απασχόλησή τους, που απαιτεί βέβαια λήψη ειδικών μέτρων. Μιλούμε για παράταση των ορίων συνταξιοδοτήσεως μιλάμε για ειδική ενίσχυση αυτών που θα μείνουν παραπάνω στην θέση εργασίας. Είναι απαραίτητο να φροντίσουμε ωστόσο με συνοδευτικά μέτρα να αποφύγουμε οποιασδήποτε επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία τους. Το εκατό των απασχολούμενων δεν έχει επαρκές εισόδημα. Η άποψή σας ως Προεδρία ποια είναι. Τι έχουν επιτευχθεί από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οδηγία για το ελάχιστο εισόδημα. Και Τελειώνω. Μία, μία φράση ακόμα κυρία Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά ε, την απόσταση μεταξύ αμοιβών γυναικών και ανδρών. Θεωρείτε ότι τα συμπεράσματα αυτά θα εγκριθούν στο Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Διότι χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, τα ίδια έχουμε. Η ίδια απόσταση παραμένει. Για Είναι πραγματικά εντυπωσιακή και η λίστα των επιτευμάτων της Βελγικής Προεδρίας. Έχετε και ένα μήνα ακόμα. Γνωρίζουμε επίσης ότι η κρίση δεν έχει παρέλθει. Οι κοινωνικές επιπτώσεις είναι σημαντικές, είναι βαριές. Πώς σχεδιάζετε να παραδώσετε την Προεδρία στους Ούγγρους γνωρίζοντας ότι η Ουγγρική Προεδρία θα κληρονομήσει μια βαριά κατάσταση, μια δύσκολη κατάσταση και πώς θα προσπαθήσετε να διασφαλίσετε ότι θα υπάρχει κάποια συνέχεια, ότι θα συνεχιστούν δηλαδή οι προσπάθειες για επίλυση όλων αυτών των πολύ σημαντικών προβλημάτων. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τηλεγραφικά γιατί δεν μένει πολλής χρόνος. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα συμπεράσματα μα που έχουν να κάνουν ε, με την μεγαλύτερη παραμονή στην εργασία των ατομών άνω των 50 και για τις πράσινες εργασίες έχουμε συγκεκριμένη αναφορά για να ζητήσουμε το Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να προσανατολιστεί για να υποστηρίξει πολύ συγκεκριμένα τις πολιτικές αυτές. Έτσι λοιπόν, ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό ό,τι αφορά την απασχόληση των ε, μεγαλύτερων σε ηλικία και την προβληματική για την επαγγελματική ε, για την υγεία στην, στο χώρο εργασίας. Ε, εδώ ε, θέλουμε όχι μόνο να διατηρήσουμε περισσότερο τα άτομα άνω των 50 στην εργασία και αυτό θα το κάνουμε με βελτίωση των συνθήκων εργασίας αλλά και με αλλαγή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας αλλά το θέμα δεν περιορίζεται στο να δούμε τι γίνεται για τα άτομα άνω των 45 ετών ε, αλλά υπάρχει άμεσο σχετισμό με, τη βέλτιστη, ε, με τις βέλτιστες προϋποθέσεις που επιτρέπουν στα άτομα αυτά να μπορέσουν να εργάζονται αρμονικά και να είναι σε δυνατότητα να συνεχίσουν για περισσότερο χρόνο την εργασία τους. Ό,τι αφορά τώρα την αδεια Φυσικά συμφωνώ απόλυτα με την απόλυτη σύνδεση ε, με την άδεια υιοθεσία ε, και ε, για την φύλαξη οι ερωτήσει που θέτουμε τη Δευτέρα, τα θέματα που θέτουμε τη Δευτέρα είναι τα πλέον επίμαχα και σας είπα ότι προσπαθούμε ε, εδώ να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για κάτι διεκτημένο, αλλά και πάλι είναι ευαίσθητα τα ζητήματα αυτά. Μας απασχολούν ιδιαίτερα τώρα. Ε, έχουμε εργαστεί εξαιρετικά υπό το τρίο και με την Ισπανική, αλλά και με την Ουγγρική Προεδρία. Συναντηθήκαμε ε, για πολλούς ε, μήνες στις Βρυξέλλες για να μπορούμε να συντονίσουμε τα προγράμματά μας, ακόμη και να αλλάζουν κυβερνήσεις, να μπορέσουμε να γνωριστούμε και να έχουμε και κοινέ κατευθυντήριε γραμμέ. Και νομίζω ότι η Ουγγρική Προεδρία είναι έτοιμη να πάρει τη σκητάλη και εμεί φυσικά είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού, όσο μπορούμε. Και για τα εθνικά σχέδια μεταρρυθμίσεων κατατίθενται με κάποιες τυχαίες προθεσμίες μπορώ να σας πω. Έτσι λοιπόν δεν γνωρίζουμε ακόμη τι περιλαμβάνουν αυτά τα διάφορα εθνικά σχέδια μεταρρυθμίσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα στο ερώτημα για ηλεκτρομαγνητικά πεδία, περιμένουμε μια πρωτοβουλία της Κομισιόν που έχει καθυστερήσει. Έτσι λοιπόν θα το χειριστεί η Ουγγρική Προεδρία. Αυτό προβλέπεται για την άδεια μητρότητας. Νομίζω ότι η προσέγγιση που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ένα συμβασμό κάποια στιγμή είναι μια προσέγγιση σε δύο χρόνους. Δηλαδή να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε για το 2020 και να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε μετά το 2020 και να δούμε πώς ε, προοδευτικά μέχρι το 2020 μπορούμε να πετύχουμε τους ε, στόχους που έχει θέσει η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 18 εβδομάδες στην αρχή, ίσως 20 ε, μετά το 2020. Δεν ξέρω, είναι κάτι προς διερεύνηση είναι ένα θέμα που πρέπει να τεθεί και να δούμε πόσο μπορούν να το δεκτούν τα κράτη-μέλη αν ε, έχουμε ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα. Ε, ίσως ε, κάποια στιγμή ε, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε όλου αυτού του δημοσιονομικού λόγου, γιατί το από το 2015 και μετά θα βρισκόμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση. Για, τις, για διακρίσεις έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε και μέσω με πρόοδο και στη στέγαση και στι χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε για του νέου. Οι ναι, είναι πραγματική προτεραιότητα. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο συζητήσαμε το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια ε, του Επίσημου Συμβουλίου του Οκτωβρίου, όπου αναλύσαμε από κοινού ποια είναι τα καλύτερα μέτρα κατά της κρίσης και για την έξοδο από την κρίση, για τους νέους που έπρεπε να διατηρηθούν και δεν θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν από τυφλέ δημοσιονομικές λογικές και ε, υιοθετήσαμε συμπεράσματα της Προεδρίας. Έχουμε διάφορες συστάσεις που συνδέονται με την έκθεση της Επιτροπής για το Youth and Move, Κινήση και αναφερόμαστε, έχουμε μία και στο Youth στην εγγύηση και απευθύνουμε και μία έκκληση να συνεχιστούν όλα αυτά από την Ουγγρική Προεδρία. Αυτές είναι οι απαντήσεις μου. Ε, Ευχαριστούμε πολύ για το το πρώτο βήμα της ανταλλαγής ε, απόψεων μεταξύ μας. Είδατε πόσο πολύ ενδιαφέρονται όλοι οι ευρωβουλευτές εδώ για τα επιτεύγματα της Βελγικής Προεδρίας. Να σας δώσω το λόγο ευθύς αμέσως. Βλέπετε, θέλουμε να συζητήσουμε για το τι μπορεί να κάνει η δικιά μας Επιτροπή για το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης. Είπατε ήδη ότι το ΕΠΣΚΟ θέλει να συμμετέχει στις συζητήσεις για την οικονομική διακυβέρνηση. Μια που είσαστε εδώ, πείτε μας πώς βλέπετε τα πράγματα και ποια είναι για σας τα σημαντικά μηνύματα. Νομίζω ότι ένα το και το ξέρουν οι συγκητέ, ότι πέρα από τη μνήμη του άρθρου 121 χρειαζόμαστε και το άρθρο 148. Πέρα όμως από αυτό το σημείο που έχει κάπως κολλήσει, για πείτε μας περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς προχωράμε. Η κυρία Μιλκέ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και να σας τα εξηγήσω καλά παρόλο που είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έχετε τρία είδη εποπτείας. Πρώτον, έχετε τη δημοσιονομική εποπτεία που έχει να κάνει με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, άρθρο 126. Ακολουθεί τη δικιά του λογική με τις νέες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας. Όχι υπερβολικά ελλείμματα, ενδεχομένω κυρώσεις κτλ. Αυτό μας απασχολεί κάπως λιγότερο, γιατί έχει να κάνει με τη δημοσιονομική πολιτική, η οποία είναι αρμοδιότητα του ΕΚΟΦΗΝ. Υπάρχει δεύτερο είδους εποπτεία, αυτή που κατά τη γνώμη μου είναι η πιο σημαντική για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την απασχόληση και εδώ είναι που θα δώσουμε μεγάλη μάχη. Και δεν είναι μάχη μεταξύ Συμβουλίου ή συσχετισμός δυνάμεων, θα ήταν ανόητο. Είναι θέμα οράματος, πώς βλέπουμε την οικονομία αγοράς και πώς βλέπουμε τη θέση της απασχόλησης και τα μέτρα για την απασχόληση που πρέπει να αποφασίζουν ε, οι Υπουργοί Απασχόληση με του κοινωνικού εταίρου και όχι μόνοι του οι Υπουργοί Οικονομικών που έχουν τη δικιά του την οικονομική λογική. Λοιπόν, μακροοικονομικό έλεγχο με νέου μηχανισμού. Εδώ προτείνεται ένας κανονισμός από την Κομισιόν. Και έχετε και την θεματική εποπτεία αυτό είναι ο τρίτος άξονας, το τρίτο σκέλος, θα μιλήσουμε λιγότερο. Είναι κλασικός ε, έλεγχος και εποπτεία που έχει να κάνει με τη στρατηγική 2020, πώς θα ελέγξουμε δηλαδή το αν πετυχαίνουμε τους στόχους μας και αν ακολουθούμε τους πέντε στόχους και τις διάφορες ναυαρχίδες που έχουμε βάλει από πλευρά ε, πρωτοβουλειών. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και μια που έχουμε λίγο χρόνο, θα επιστήσω την προσοχή σας στη νέα λογική της μακροοικονομικής εποπτείας. Πώς την έχουμε συλλάβει όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Εδώ μπορούμε να προχωρήσουμε σε καινοτομίες, τηρώντας όμως πλήρως το άρθρο 148. Βλέπετε, προβλέπετε τον Ιανουάριο να κατατεθεί μια κοινή έκθεση για την οικονομική κατάσταση, Joint Survey Report, που εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας εισαγάγει σε όλη αυτή τη διαδικασία μακροοικονομικής ε, εποπτείας. Στη συνέχεια έχετε συστάσεις που πρέπει να υιοθετηθούν από το Εαρινό Συμβούλιο. Προκειμένου οι συστάσεις αυτές να υιοθετηθούν και απευθύνονται στα κράτη-μέλη, έτσι εν ώψη των ε, δικών τους προγραμμάτων ε, μεταρρύθμισης. Φτάνουμε, βλέπετε, σε ένα περίοδο που η Ευρώπη έχει μεγαλύτερο βάρος. Προηγουμένως, λοιπόν, θα έπρεπε να έχουν υπάρξει συστάσεις που να έχουν προετοιμαστεί από το Συμβούλιο Κοφίν για τα μακροοικονομικά ζητήματα και όταν αναλύεται την επιστολή του Επιτρόπου ή τις διάφορες άλλες αναλύσεις, όταν μιλάμε για μακροοικονομική πολιτική, το 70% έχει να κάνει με την απασχόληση. Είναι ποιο είναι το κόστος της εργασίας, φορολόγηση της εργασίας ή των μισθών, είναι εδώ η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, οι δεξιότητες, τα προσόντα που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα. Είναι τα θέματα καμψίας στην αγορά εργασίας κλπ. Άρα λοιπόν αυτό που διακυδεύεται σε αυτό το στάδιο είναι αν για το Ερεινό Συμβούλιο αφήσουμε μόνο το Συμβούλιο Κοφίν να κάνει συστάσεις ώστε να ετοιμαστεί το σύνολο των συστάσεων στη συνέχεια για τις ε, χώρες μέλη, προκειμένου να ετοιμάσουν τα εθνικά τους ε, προγράμματα, χάσαμε. Γιατί οι πιο αρμόδιοι σε θέματα απασχόλησης, οι υπουργοί απασχόλησης, δεν θα μπορέσουν να επηρεάσουν και να βάλουν τη δικιά τους νότα στις συστάσεις αυτές. Γι' αυτό προτείνουμε οι συστάσεις που γίνονται και πάνε στο Ερηνό Συμβούλιο να γίνεται και από το ΕΚΟΦΗΝ, που έχει βέβαια το δικό του ρόλο, πολύ ενδιαφέροντα, αλλά και από ε, το ΕΠΣΚΟ. Εγώ τουλάχιστον έτσι θα ήθελα να το οργανώσω και αυτό προτείναμε, αφού έχουμε συζητήσει και θα συζητήσουμε κι άλλο και με σας και με τους κοινωνικούς εταίρους για να φτάσουμε σε προτάσεις βάση το 148 εκ παραλίλου και ίσως και σε συνεργασία, με συντονισμό με το Συμβούλιο, με το ΕΚΟΦΗΝ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Αυτό είναι το πρώτο που λέει το άρθρο 148. Είναι απόλυτα λογικό βάσει της νέας διάστασης. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι επιμονή μου βάσεως, οπότε είναι νέα μηνύματα που βάζουμε. Την ίδια ορολογία χρησιμοποιεί και το ECOFIN. Αν αυτοί μπορούν να κάνουν key messages, όπως τα λέει η ορολογία τους, μπορούμε και εμείς. Μετά το Πάσχα, λοιπόν, θα έχουμε τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης βάσει των συστάσεων αυτών. Μετά θα υπάρξει ένας δεύτερος γύρος που είναι οι συστάσεις αναχώρα. Και αυτό το προβλέπει το άρθρο 148 σε ένα από τα τελευταία εδάφια που είναι μεν σε εθελοντική βάση, αλλά μπορούμε να το κάνουμε συστηματικά κάθε χρόνο. Μετά την ανάλυση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης, που την ανάλυση την κάνει η Κομισιόν, θα έπρεπε εμείς όπως και το κοφίν, έτσι και εμείς να κάνουμε προτάσεις αναχώρα, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι και αναχώρα μπορούμε να έχουμε τις πιο καλές συστάσεις. Μην αφήσουμε πάλι μόνο τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν ε, συστάσεις για την απασχόληση και οι συνάδελφοι από την απασχόληση να μην έχουν ε, λόγο επ' αυτού. Το άρθρο 148 λοιπόν μπορεί κάλλιστα να είναι η νομική βάση η οποία θα μας επιτρέψει πριν από το Συμβούλιο του Ιουνίου βάσει των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης να κάνουμε εμείς προτάσεις για την απασχόληση. Και έτσι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γίνουν οι προτάσεις χώρα και από τη δικιά μας την πλευρά και από το ΕΚΟΦΗΝ. Σε συντονισμό μεταξύ μας, ελπίζω. Αυτό διεπιδεύεται λοιπόν. Αν διαβάσετε τον κανονισμό για την μακροοικονομική διακυβέρνηση, δεν υπάρχει μνήμα στο άρθρο 148. Οπότε κινδυνεύουμε να μην τηρηθεί καθόλου. Εδώ προσπαθούμε να κάνουμε μία επανάσταση, ενώ το ΕΚΟΦΗΝ φαίνεται να είναι ο μόνος συνομιλητής με τα διάφορα υποσυμβούλια του και εμείς δεν υπάρχουμε πουθενά. Είναι λάθος αυτός ο δρόμος. Πρέπει να υπάρχει πολιτική ισορροπία. Και για να είναι πιο αποτελεσματική η πολιτική απασχόληση πρέπει να είναι αλλιώ τα πράγματα. Την πολιτική για την απασχόληση πρέπει να την κάνουν οι υπουργοί οι οποίοι θα πρέπει και να εφαρμόσουν τη σχετική μεταρρύθμιση. Δεν είναι οι υπουργοί οικονομικών που θα μας πούνε τι πρέπει να κάνουμε στην υγεία. Να, ένα άλλο θέμα. Ή για τις συντάξεις. Και οι υπεύθυνοι να πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα που υιοθετηθούν χωρίς προηγουμένως να έχουν πει τη γνώμη τους, δεν είναι αποτελεσματικό κάτι τέτοιο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε τη συμμετοχή την δικιά μας σε αυτά τα θέματα. Στα συμπεράσματα έψκο του Οκτωβρίου το είπαμε ξεκάθαρα. Υπάρχει και στις κατευθυντήριες γραμμές. Και πετύχαμε τη μικρή αυτή μνήμα που έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τέλειο Οκτωβρίου. Ένα από τα πράγματα που διακυδεύονται με τον προσιοθέτηση κανονισμού είναι να λαμβάνετε υπόψη το άρθρο 148 και λαμβανόμαστε και εμείς υπόψικη. Πρέπει αφενός να έχουμε αποτελέσματα και δεύτερον να διαθέτουμε, τα... να διαθέτουμε αποτελεσματικά όργανα. Η επανάσταση που προσπαθήσαμε να κάνουμε και την κάναμε είναι ζητήσαμε από την Επιτροπή για την Απασχόληση, την ΕΜΚΟ, και εμείς αυτό το εγκρίνουμε για να μια που γνωρίζουμε και την μακροοικονομία και την απασχόληση, δεν έχει κανείς να μας δώσει μαθήματα. Αυτό λοιπόν που ετοίμασε αυτή η Επιτροπή και που θα υιοθετήσουμε εμείς τη Δευτέρα είναι το Joint Assessment ε, Report. Πρόκειται για μια έκθεση αξιολόγησης που αναλύει τις αγορές απασχόλησης και θα είναι κάτι σαν βαθμολόγιο ή τέλος πάντων σαν οδικός χάρτης για να βλέπουμε ποια είναι η εξέλιξη των αγορών απασχόλησης, τι γίνεται με την ανταγωνιστικότητα, με την κατάρτιση. Εκεί συμπεριλαμβάνεται η προβληματική απασχόληση ευρύτερα και όχι όπως παλιότερα από τους δείχτες μόνο οι μισθοί αναφέρονταν. Φυσικά και πρέπει να μιλήσουμε και για τους μισθούς, αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος δείχτης. Προβλέψαμε λοιπόν αυτό το μέσο για να αναλύουμε συνεχούς βάσεως το κατά πόσο τηρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές στα πλαίσια της νέας ε, οικονομικής διακυβέρνησης και για να μπορούμε να την ε, αναλύουμε. Έτσι ώστε η ανάλυση μας να είναι περισσότερο στο βάθος και να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται στις αγορές απασχόλησης. Αυτά θα εγκρίνουμε τη Δευτέρα. Προβλέπεται και έλεγχος της απασχόλησης γενικότερα με όλους τους δείκτες και επιμέρους δείκτες. Αυτό είναι ένα από τα κύρια θέματα. Η συζήτηση θα κρατήσει βέβαια πριν ε, εγκριθούν ε, τα πάντα. Εμείς όμως θα επιμείνουμε. Και πριν τον Ιανουάριο θα υπάρχει η κοινή έκθεση της Επιτροπής και ευχαριστώ και την Ουγγρική Προεδρία η οποία στο δικό της χρονοδιάγραμμα έχει ήδη συμπεριλάβει το δικό μας τρόπο εργασίας προκειμένου να καταλήξουμε σε συστάσεις για τα νέα μέσα διακυβέρνησης που θέλουμε να περάσουν στο Εαρινό Συμβούλιο για να γίνουν εν ώψη του Συμβουλίου του Ιουνίου και η αναχώρα εκθέσεις. Είπαμε για νομική βάση χρησιμοποιούμε το 148. Το Κοινοβούλιο έχει πάντα τη θέση του, εγώ άλλο που δεν θέλω να ενισχύεται περισσότερο και υπάρχει βέβαια και θέση συζήτηση αυτή και για τους κοινωνικούς εταίρους. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη συζήτησή μας και πιστεύω ότι θέλουμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Η δέσμευση αυτής της Επιτροπής είναι επίσης σημαντική. Ως εισηγήτρια του ίμιση του πακέτου, το άλλο μισό το έχει αναλάβει ο συναδελφός Δαβίτ Καζάκη που θα έλθει εδώ σε λίγο. Ε, θα ήθελα να επανέλθω σε δύο-τρία σημεία. Καταρχήν, ε, σε ό,τι αφορά τα ε, κείμενα που έχουμε πει και συζητούμε, μας αναφέρατε συγκεκριμένα δύο. τα τελευταία αφαιρούν περισσότερα την μακροοικονομική υποπτία. Αλλά προς στιγμή κανένα από τα κείμενα αυτά δεν συμπεριλαμβάνει τη δυναμική του Ευρωπαϊκού Ξαμήνου ω τέτοια. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αυτά για να εντάξει αυτή τη δυναμική του Ευρωπαϊκού Ξαμήνου. Και καθώς ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν μεταφράζεται, στην πραγματικότητα των κειμένων αυτών, τα εργαλεία που έχει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διάθεσή του δηλαδή όσα προϋπήρχαν ε, πριν από τη μεταρρύθμιση αυτή και όσα υπάρχουν σήμερα, φαίνεται να εξαφανίζονται στην άμμο. Και σε ό,τι αφορά ζητήματα απασχόληση, εγώ δεν θα ήθελα εξαιρετική δουλειά που κάναμε με βάση την έκθεση Τσαβάουρη για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση να εξαφανιστούν. Δηλαδή δεν υπάρχουν πια, κανένα δεν μιλάει για αυτού του μεγάλου προσανατολισμού που συζητούμε εδώ και για τι κατευθυντήριε γραμμέ για την απασχόληση. Ενώ πρόκειται για εργαλεία που αναφέρουν τη συνθήκη και τα οποία ενημερώνεται ή ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι σημασία λοιπόν πρέπει να δώσουμε σε αυτά τα εργαλεία. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα επανεισαγάγουμε στο κείμενο ή αν όχι, ε, με τι θα αντικαθιστούμε Δηλαδή έχουμε τελείως χαλαρές διαδικασίες. Είναι πραγματικά δύσκολη ε, η κατάσταση αυτή. Η τρίτη μου παρατήρηση έχει να κάνει με το scoreboard, το βαθμολόγιο. Γιατί είπατε πώς κινητοποιήθηκε για να καταστήσει επαγγελματική τη διαδικασία και τους δείκτες ε, για να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς. Και φυσικά και όσοι ασχολούνται με τις κοινωνικέ υποθέσει πρέπει να είναι οι καλύτεροι. Ε, και έχετε δίκιο ότι ήταν ε, αυτή ε, μια προσδοκία και ίσως θα αποτελέσει πλεονέκτημα για τι διαπραγματεύσει. Όμω, αν δούμε τι προβλέπετε σήμερα στα κείμενα με τα οποία ασχοληθήκαμε, στο scoreboard δεν υπάρχει τίποτα σήμερα. Δεν υπάρχει καμία ε, ένδειξη. Ακούσαμε ότι η Επιτροπή θα το κάνει, αλλά πώς θα το κάνει η Επιτροπή και τι πρέπει να βάλουμε μέσα. Εγώ νομίζω ότι εδώ εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσουμε λεπτομερώς ε, ε, για το τι θέλουμε να συμπεριλαμβάνεται στους δείκτες. Δεν είμαστε εμπειρογνώμονες στους δείκτες, αλλά αν είχαμε και τη δική σας άποψη χρήσιμη θα ήταν. Και κάτι ακόμη για το θέμα των κυρώσεων. Φυσικά περισσότερο αυτό είναι αρμοδιότητα του ΕΚΟΦΗΝ ή της ΕΚΟΝ, αλλά θα έχει και κοινωνικές επιπτώσεις. Ε, έτσι λοιπόν, εδώ έχετε να διαβάσετε ένα μήνυμα ή ε, θεωρείτε ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί σε άλλα βήματα και ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε εμείς καθόλου το ζήτημα αυτό. Καθώς έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, θα δώσω αμέσως το λόγο στους συναδέλφους που θα ήθελαν να τοποθετηθούν. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν πρόσθετες ερωτήσεις για το σημείο αυτό. Μάλιστα, σας ξαναδίνω το λόγο λοιπόν. Μάλιστα. Κοιτάξτε, οι ερωτήσεις σας ε, είναι πραγματικά πολύ στοχευμένε, γιατί μιλήσαμε για το Ευρωπαϊκό Ξάμεινο, δεν υπάρχει στον κανονισμό, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη η οδή για τη λήψη απόφαση. Έχουμε το Χερμαυροβέο που ασχολείται με την Task Force, ε, όπου υιοθετείται και τα συμπεράσματα και δεν ε, εφαρμόζεται εκεί, δεν ισχύει το άρθρο 148, αλλά έμεσα και ταυτόχρονα έχουμε ε, και την Επιτροπή πριν που έρχεται να επισέλθει εδώ πριν να υιοθετηθεί η έκθεση της Tax Force. Ε, πάντως, ε, για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, εγώ νομίζω στις συζητήσεις που θα κάνετε για τον κανονισμό, επί της ουσίας, το μόνο επίσημο έγγραφο που μιλάμε για το θέμα αυτό και εξηγούμε το, χρονικά στάδια είναι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου έψικο του Οκτωβρίου στο οποίο γίνεται μνήα στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί ε, αναφέρονται ε, οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε βήμα του Συμβουλίου και σε κάθε σχηματισμό του Συμβουλίου. Ίσως ε, τώρα αυτό θα μπορούσατε να εντάξετε ε, είτε σε αυτό το μέσο είτε σε κάποιο άλλο. Αλλά σίγουρα θα έπρεπε να ενταχθούν. Αυτό εσείς θα το αποφασίσετε βέβαια το πού. Γιατί το χρονοδιάγραμμα είναι σημαντικό και πρέπει να δούμε και πώς συμπεριλαμβάνουμε και τις νομικές βάσεις 121-148. Τώρα η ρωτή σας για το scoreboard, για το βαθμολόγιο είναι ιδιαίτερα στοχευμένη και είναι συζήτηση που πρέπει να γίνει τώρα, γιατί μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει ολοκληρωθεί, ούτε έχει καταγραφεί. Η Κομισιόν ε, σε αυτούς τους ε, διάσημους δείκτες που είναι οι μόνοι για τους οποίους κάνουμε λόγο σήμερα και που στο στάδιο αυτό είναι η υποποκλειστική διαχείριση του ΕΚΟΦΗΝ, ε, είναι τα ενεργητικά στο εξωτερικό για την ανταγωνιστικότητα, είναι το κόστος των μισθών, είναι το μόνο στοιχείο για την απασχόληση και δεν αρκεί φυσικά. Έχουμε τη χρέωση, τη στέγαση, ε, το χρέος υπό το, τις κατασκευαστικές εργασίες κτλ. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε πώς οι δείκτες ε, πώς τους δείκτες αυτού προσθέτουμε, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε και 25, πώς προσθέτουμε λοιπόν κάποιους άλλους δείκτες. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση επί των μισθών και πρέπει να σεβαστούμε και το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και τις εθνικές διαδικασίες. Δεν όμως ε, ένας, ε, ένα δείκτη ε, που να, έχει, να κάνει με την απασχόληση δεν μπορούμε να μην το φανταστούμε. Έτσι λοιπόν, ένα σύνολο δικτών προβλέπονται από την Επιτροπή Απασχόλησης. Μιλάμε για σημαντική στοιχεία, αλλά για μένα τα πιο σημαντικά είναι, παραδείγματο χάρη, το ποσοστό τη απασχόληση ε, και κάτι που έχει να κάνει με την παραγωγικότητα και για τι συμπληρωματικέ πτυχέ, έτσι ώστε να υπάρχει ένα σύνδεσμο μεταξύ ε, των δύο αυτών σχηματισμών, να γίνει μια αναφορά στο Joint Assessment Framework, ε, σε αυτό το πλαίσιο το οποίο καλύπτει το σύνολο των δικτών ε, απασχόλησης για να εμβαθύνουμε στην ανάλυση. Εγώ μπορώ να φανταστώ να πάρουμε κάποιους κύριους δείκτες, αλλά ε, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και κάποιους πιο συγκεκριμένους δείκτες, αλλά για την απασχόληση θα μπορούσαμε να έχουμε μία πιο στοχευμένη και συγκεκριμένη ανάλυση βάσει των εργασιών της ΕΜΚΟ. Σε ό,τι αφορά τις αυτή είναι μια πολιτική συζήτηση πιο ευρεία από αυτή που διεξάγει το Συμβούλιο, αλλά φαίνεται πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν όλοι οι πρωταγωνιστές, γιατί όταν μιλάμε για μακροοικονομική εποπτεία, όταν έχουμε μια πραγματική ανισορροπία, φτάνουμε στη σημερινή κατάσταση, δηλαδή να μπορούμε να ε, έχουμε κάποια στιγμή κυρώσεις 0,1 του ΕΠΑ ε, ανακρατοσμέλος 0,2 είναι για το περιβολικό έλλειμμα και για το σύμφωνο σταθερότητα, ενώ όταν ε, είμαστε στο πλαίσιο της μικροοικονομικής εποπτείας έχουμε κάτι όχι τόσο κακό, 0,1. Έτσι λοιπόν, ε, πώς να αφήσουμε στα ίδια χέρια τόσο μονόπλευρες αποκλειστικέ αναλύσει και την επιλογή των κυρώσεων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό τουλάχιστον οι αναλύσεις των ισορροπιών και οι συστάσεις ε, να αναλυφθούν από διάφορους ακόμη και αν το άρθρο 148 δεν επιτρέπει τις κυρώσεις. Ε, τουλάχιστον όμως ε, θα πρέπει να έχουμε πολλαπλές αναλύσεις και φυσικά και το Κοινοβούλιο και οι κοινωνικοί εταιροί πρέπει να συμμετάσχουν και για τις κατευθυντήρες γραμμές για την απασχόληση. Όταν μιλώ για το ευρωπαϊκό εξάμεινο και για τη σημασία να μπορούμε να συμπεριλάβουμε και αυτή τη λογική σε ένα από τους δύο κανονισμούς. Το λέω αυτό προκειμένου να έχουμε συνέπεια στο πώς εφαρμόζουμε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και το 148 σε αυτή την θεματική. Γιατί για αρκετό καιρό είχαμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι όταν μιλάμε ε, για τις κατευθυντήριες γραμμές υπό το 148 ε, ουσιαστικά εδώ συμπίπτουμε με την ερμηνεία του κοφίν, αλλά πρέπει να υπάρχει και μνήμα στον κανονισμό. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Υπουργέ για αυτή τη συνεργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Βελικής Προεδρίας που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη κάθε επιτυχία για το τελευταίο ΕΦΣΚΟ και εξ ονόματος όλων των συναδέλφων μπορώ να σας πω αν και το ξέρετε ότι εκτιμήσαμε πάρα πολύ τη συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστούμε.

Chers Α συνεχίσουμε τις εργασίες μας, ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτσι με το υπαριθμόν πέντε θέμα της ημερήσιας διάταξής μας θα φτάσουμε στην εξέταση των τροπολογιών στην ε, γνωμοδότηση της κυρίας Παπαδοπούλου σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων 2007 έως 2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Κυρία Σιγήτη, έχετε το λόγο. Mrs. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συνολικά 59 τροπολογίες κατατέθηκαν στην ε, γνωμοδότησή μου. Μεταξύ αυτών των 59 τροπολογιών 27 ε, συγχωνεύτηκαν σε 6 συμβαστικές τροπολογίες που θα ψηφιστούν και οι υπόλοιπες ατομικά. Εγώ θεωρώ ότι είναι βέβαια βελτίωση, διότι με τις συμβαστικές τροπολογίες μπορέσαμε να πάρουμε να περιλάβουμε τις περισσότερες από τις ιδέες που υπέβαλαν οι συναδελφοί μου. Μόνο για τρεις τροπολογίες έχω κάποιους δισταγμούς σχετικά με το αν θα έπρεπε να τις περιλάβω ή όχι. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων μου, αφού βεβαίως ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι συνεργάστηκαν και μου φαίνεται πως υπάρχει και συμβιβασμός, ίσως με εξαίρεση μιας πολιτικής ομάδας που φαίνεται δεν θέλει να τον υπερψηφίσει. Ελπίζω βέβαια στο τέλος της συζητήσεως όλοι να συμφωνήσουμε και να μπορέσουμε να περιλάβουμε όλες τις τροπολογίες στην γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Επιθυμεί κανείς να παρέμβει. Thank you, madam. Ε, Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λέει η κυρία Χάρκιν. Η κυρία Καστανόβα δεν είναι σήμερα παρούσα και μιλώ εκ μέρους της. Συμφωνεί με τις συμβιβαστικές τροπολογίες ένα ή δύο σχόλια μόνο για ορισμένες άλλες τροπολογίες. Δικό μου σχόλιο αναφέρεται στο 30 της κυρίας Φιγκερέντο που ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νέα πρωτοβουλία για αναθεώρηση των κριτηρίων της συγχρηματοδότησης. Η δική μου άποψη είναι ότι όντως χρειάζεται να το εξετάσουμε αυτό γιατί οι πιο πρόσφατες εκθέσεις μας λένε ότι μόνο 10% από τα 374 εκατομμύρια που έχουν διατεθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί. Και ένας από τους λόγους, και υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι, είναι ότι οι εθνικές κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις των χωρών μελών δηλαδή, που δεν έχουν <clears throat> πλέον ρευστό, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα έργα. Επίσης η τροπολογία 19 της κυρίας Σρέντερ. Εδώ έχω μία ερώτηση. Όταν λέτε για μεταφορά πόρων από το ESF στο ERDF, ε, ε, ε, εμείς διαφωνούμε διότι δεν είναι προφανής η ορατότητα. Αλλά ήταν επαρκείς αυτές οι μεταφορές πόρων και γιατί έγιναν. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει κυρία Γιάσλοβιέτσκα. Ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια που με τόσο ανοιχτό πνεύμα εκπώνησε το τελικό κείμενο συμβιβασμών και τονίζω επίσης ότι από τις έξι συμβιβαστικές τροπολογίες εμείς υποστηρίζουμε τις πέντε. Δεν υποστηρίζουμε μία από αυτές, μία από τις έξι. Δεν μπορέσαμε να βρούμε συμφωνία δηλαδή σε αυτήν την υπαριθμόν πέντε και δεν μπορέσαμε να βρούμε συμφωνία, να καταλήξουμε συμφωνία για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ήδη στην εισαγωγή γίνεται αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσα στα πλαίσια της καταπολεμής της στόχιας. Όμως το Ταμείο αυτό έχει ως στόχο να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, να ε, ενισχύσει το επιχειρήν, να ε, χρηματοδοτήσει μετεκπαιδευτικά προγράμματα. Βέβαια η καταπολέμηση της φτώχειας είναι σημαντική, αλλά ξεφεύγει από τον στόχο του προγράμματος αυτού, του ταμείου αυτού. Που έχει στόχο να κινητοποιήσει την αγορά εργασίας. Πάλι για την 5 δεν συμφωνούμε με την οικονομική αυτονομία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η πολιτική συνοχή είναι μια πολιτική που βασίζεται σε ένα κοινό προπολογισμό. Ε, δεν επιθυμούμε να διαρρεθούν οι προπολογισμοί. Πριν από μήνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο ψηφίσματα όπου ολόκληρο το Κοινοβούλιο ψήφισε κατά της άρσης αυτής της αυτονομίας. Και αναφέρομαι ειδικά στο ψήφισμα για την πολιτική συνοχής και το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτά είναι βέβαια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να δεχθούμε και γι' αυτό δεν μπορέσαμε να υπερψηφίσουμε την ε, συμβαστική αυτή τροπολογία. Υποστηρίζω και ορισμένε από τις ε, τροπολογίε που κατατέθηκαν με στόχο να αυξηθεί η αποδοτικότητα του Ταμείου, να αυξηθεί δηλαδή η χρηματοδότηση ε, προγραμμάτων διαβίου κατάρτισης και όλων αυτών των ε, προγραμμάτων που διευκολύνουν την επιστροφή στην επαγγελματική ε, δραστηριότητα. Λούντβιξον. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, ζητώ συγγνώμη, λέει ο στο 6 δεν έχουμε φτάσει. Α, όχι, όχι, όχι, δεν είμαστε στο 6. Η κυρία Σρέντερ. Πρώτα θα ήθελα να απαντήσω την κυρία Χάρκιν. Δεν έχω ε, κοιτάξει το αγγλικό κείμενο, διότι υπέβαλα τα κείμενά μου στα γερμανικά, αλλά θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο ε, ζητούμε αυτά που ζητούμε. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια το ποσοστό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μέσα στα λειτουργικά προγράμματα έχει μειωθεί, έχει γίνει μικρότερο, διότι οι χώρες μέλη έχουν εθνικούς πλέον envelopes, φακέλους και αποφασίζουν πόσα θα δώσουν για το ένα ταμείο και πόσα για το άλλο. Και το ποσοστό του ταμείου αυτού μειώνεται. Εκεί νομίζω λοιπόν πρέπει να προσέξουμε να μην μειωθεί κι άλλο, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ωστόσο σημαντικό εργαλείο για την πολιτική της απασχόλησης. Και αυτό συνδυάζεται και με τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις, δηλαδή πόσο ξεκάθαρο είναι το περιεχόμενο του κανονισμού. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω την ανάλυση αυτή, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδια δεν την έχει κάνει την ανάλυση αυτή. Η Πρόεδρος επιθυμεί, κανείς άλλος, παρακαλώ κυρία Συγκήτρια. Θα σχολιάσω τις τρεις αυτές παρεμβάσεις. Πρώτα, για την 30 της κυρίας Φιγκερέντο. Εγώ προσωπικά την δέχομαι την τροπολογία που νομίζω ότι η σύστασή της είναι καλή. Δηλαδή, να προχωρήσει μια πρωτοβουλία για την επανεξέταση των κριτηρίων συγχρηματοδότησης από πλευρά των χωρών μελών ώστε να μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν και χώρες οι οποίες έχουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσχέρειες. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανέ. να εφαρμοστεί στην πράξη δηλαδή. Για την 19 τώρα, τροπολογία 19 της κυρίας Σρόιντερ και για τον ίδιο λόγο που ε, μίλησε η κυρία Χάρκιν, δεν είμαι βέβαια πώς αιτιολογείτε την στάση σας, την θέση σας μάλλον, ότι έχει μειωθεί δηλαδή το ποσοστό του ταμείου αυτού μέσα στα παρελθόντα χρόνια. Νομίζω ότι δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε κάθε βέβαια επιμέρους χώρα. Όπως είναι γραμμένο πάντως, εμείς δεν θέλουμε να μειωθεί το ταμείο αυτό υπέρ άλλων ταμείων όπως ε, του Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δηλαδή επί της ουσίας συμφωνώ με την θέση σας αυτή. Αλλά η ερώτησή μου είναι πώς την στηρίζετε την άποψη αυτή. Δεν γνωρίζω αν έχετε ίσως κάποια έξτρα στατιστικά δεδομένα που μπορούν να στηρίξουν τον ισχυρισμό αυτό. Γι' αυτό το λόγο ε, πρότεινα εγώ στη λίστα ψηφοφορία αποχή. Γιατί δεν έχω δει δεδομένα στοιχεία πώ υποστηρίζετε την, απο... την άποψη. Επί τη ουσία του αιτήματο συμφωνώ να μην μειωθεί. Αλλά πώ πώς το ε, θεμελιώνεται τον ισχυρισμό αυτό. Τώρα για τον συμβιβασμό. Μιλήσαμε με την Τανούτα και για όλα τα θέματα που έχετε υποβάλει. Η συμβιβαστική ε υπάρχει μια διαφορά στην προσέγγιση. Σε τρία σημεία δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε. Πρώτο, κατά τη γνώμη, μου, είναι ότι το κοινωνικό ταμείο είναι βασικό εργαλείο το οποίο έχει ως στόχο την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση όμως και της στόχιας, την καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και των κοινωνικών διακρίσεων κατά ανθρώπων με ε, αναπηρίες, ε, μεταναστών κλπ. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό, διότι κάποιο ζήτησε να διαγραφεί η παράγραφος αυτή και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας. Αυτό ήταν ένας από τους λόγους για, τον οποίο, για τους οποίους δεν συμφωνήσαμε τελικά. Το δεύτερο ήταν για την οικονομική αυτονομία. Νομίζω ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να διαθέτει χρηματοδοτική αυτονομία και εδώ υπήρξε μια δεύτερη διαφωνία. Επίσης και λίγο παρακάτω, μετά από την συζήτηση κατέστη σαφές ότι δεν μπορούσαμε να συμβιβαστούμε. Δεν ξέρω αν ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα το υποστηρίξει αυτό ή όχι. Η δική μου ελπίδα είναι να λάβουν υπόψη τους το ότι ένας από τους στόχους της Ευρώπης 2020 είναι η καταπολέμηση της φτώχειας ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και κοινωνικού αποκλεισμού και να δοθεί κάποια χρηματοδότηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι άλλες τροπολογίες, κατά τη γνώμη μου, είναι αποδεκτές, όλες τους. Οι μόνες τρεις ήταν οι παριθμών 13, 19 και η συμβαστική ε. Όλες τις υπόλοιπες τις δέχομαι. Ε, θέλετε να ανοίξετε ξανά την συζήτηση. Μα νόμιζω ότι συζητήθηκαν όλα. Όλοι μπόρεσαν να τοποθετηθούν. Παρακαλώ κύριε Ιουζεύσκα. Ευχαριστώ. Θέλω να σχολιάσω τις παρατηρήσεις της εισηγήτριας, επιτρέψτε μου, όσον αφορά την μείωση της ένδυας, που αποτελεί την ε, βάση, μιλάει και για την ισότητα εκεί, αυτό λέει ο συμβιβασμό. Δεν μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε έτσι όπως διατυπώνεται. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια συνοχή στη διατύπωσή μας και να υπάρχει συνοχή με ό,τι έχουμε εγκρίνει προηγουμένω. Το ίδιο ισχύει και για την οικονομική ανεξαρτησία. Πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες, εγκρίναμε ένα ψήφισμα όπου όλοι συμφωνήσαμε να απομακρυνθούμε από την διάταξη αυτή. Γιατί τελικά αυτοί που διαβάζουν από τους πολίτες τα έγγραφά μας, τι θα πούνε, ότι το αναζητάμε ζητάμε στο ένα έγγραφο και κάτι άλλο ζητάμε σε άλλο έγγραφο. Πρόεδρος. Ωραία, κύριε Σόντερ και εσείς. Ξανακοίταξα το αγγλικό. Το αγγλικό λοιπόν είναι εντάξει το κείμενο. Αυτό εννοώ και εγώ λέει στο αγγλικό κείμενο ότι οι χώρες μέλη αποφασίζουν πόσα λαμβάνει το ένα ταμείο και πόσο, πόσα το άλλο όταν αναπτύσσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα. Και εξετάζοντας όλες τις χρηματοδοτικές περιόδους, και για μένα είναι η τρίτη αυτή, βλέπει κανείς ότι το κοινωνικό ταμείο έχει μειωθεί ποσοστία. Και αυτό που θεωρώ εγώ είναι ότι πρέπει να καθίσουμε να το σκεφτούμε αν πράγματι είναι καλό αυτό. Ωραία, δεν νομίζω ότι χρειάζονται άλλα σχόλια. Η ψηφοφορία για την έκθεση αυτή θα γίνει εδώ αύριο επί της ουσίας ε, επιτροπή, η περιφερειακή, θα ψηφίσει στις 26 Ιανουαρίου. Έχει καιρό δηλαδή για να λάβει υπόψη της και τις δικές μας προτάσεις. Φτάνουμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Όλε Λούντβικσον για να μας ε, παρουσιάσει την γνωμοδότησή του που απευθύνεται στην Επιτροπή Ήτρε Βιομηχανίας και έχει να κάνει με το εξή θέμα, μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο για να μας μιλήσετε για τις τροπολογίες που έχουν ε, κατατεθεί, αλλά και για τις τέσσερις συμβιβαστικές Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές από τις άλλες πολιτικές ομάδες για την εξαιρετική συνεργασία. Συμφωνήσαμε επί τέσσερις συμβιβαστικές τροπολογίες. Από τις έξι παραγράφους οι τέσσερις έτυχαν συμβιβασμού που από ό,τι φαίνεται μπορεί να είναι να αποτελέσουν λύσεις. Έτσι λοιπόν με τις τροπολογίες ε, που παρουσιάστηκαν μπορούσαμε να βελτιώσουμε το κείμενο κυρίως ε, σε ό,τι αφορά την ε, κατάρτιση, της κοινωνικής σχέσης και νομίζω ότι έχουν παραμείνει και κάποια επίμαχα στοιχεία Ίσως ε, θα ήταν ε, χρήσιμο να υπάρχει και κάποια περαιτέρω ε, διόρθωση. Πάντως σας ευχαριστώ για το λόγο και ελπίζω να μπορέσει να εγκριθεί αυτή η γνωμοδότηση. Υπάρχουν αντιδράσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Χάρκιν. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κυρία Χασπανόβα που είπατε δεν ήταν εδώ. Από ό,τι φαίνεται δεν βλέπω πολύ καλά. Μάλλον ε, το ίδιο συμβαίνει και με το μυαλό μου. Πάντως ζητώ συγγνώμη, αλλά ο κ. Κρέτσμαν δεν είναι εδώ και μου ζήτησε να κάνω κάποια σχόλια εξ ονοματός του. Είπε ότι θα ήθελε μια βιομηχανική πολιτική που να αναγκαλίζει την ε, ε, οικονομία της αγοράς, αλλά θα ήθελε να προωθεί και τη δυνατότητα των εταιριών να υλοποιούν επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Θα πρέπει να ε, μπορούν να αποφασίζουν ποιες είναι οι τεχνολογίες του μέλλοντος. Οι αγορές όμως προσφέρουν τους κατάλληλους πόρους για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο της όλης αλυσίδας ε, εφοδιασμού προκειμένου να ληφθούν υπόψη και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει ε, να ε, κατανοήσουν καλύτερα τα ωφέλη της διασυνορικής συνεργασίας και ένας αριθμός τέτοιων εταιριών πρέπει να επωφεληθούν από ασφαλή χρηματοδότηση και επίσης θέλει να τονίσει ότι οι κοινωνικοί εταίροι είναι σε καλύτερη θέση για να διαχειριστούν τις κατάλληλες ε, προσαρμογές ε, κατόπιν της οικονομικής κρίσης. Όμως πιστεύει ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών να μετριάσουν ε, τα κοινωνικά προβλήματα και να διασφαλίσουν τα προσόντα των εργαζομένων. Η διαβίου μάθηση και κατάρτιση είναι σημαντικές σε αυτό το πλαίσιο και σε ό,τι αφορά τη συμβαστική τροπολογία Β θεωρεί ότι η φράση και νέες τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της παροχής ενέργειας και της μείωσης ε, των εκπομπών του δεξιού του άνθρακα ενώ ε, φυσικά υποστηρίζει την εξέβρεση τέτοιων λύσεων θεωρεί ότι είναι κάπως στενό να χρησιμοποιήσουμε μόνο τους δύο τομείς στην παροχή ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών και προτιμά μια πιο γενική προσέγγιση αλλά θεωρεί ότι καλό είναι να συζητηθεί αυτό περαιτέρω με τον συγητή. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που να ζητά το λόγο. Ο κύριος Λούντβικσον, θέλετε να αντιδράσετε. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Κοιτάξτε, να δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. είχαν ε, σταλεί αυτές οι προτάσεις, ε, παρ' όλα αυτά και όλοι είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν. Δεν υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ε, βέβαια, εγώ όσα υπόθηκα φυσικά και θα τα λάβω υπόψη. Σας ευχαριστώ. Bon, καλώ. Euh, Πρόεδρος, καλώς. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει συμφωνία για τους τέσσερις συμβιβασμούς. Θα ψηφίσουμε αύριο και 13 Ιανουαρίου θα ψηφίσει Ήτρε. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο 8. Εδώ θα εξετάσουμε τις 82 τροπολογίες... Α, συγγνώμη λέει η Πρόεδρος. Πού θέλει να παρέμβει η Επιτροπή? Σε ποιο σημείο? Α, ωραία. Σημείο 7. Ευχαριστώ που μας επιτρέπετε να πάρουμε το λόγο. Είμαστε από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεις και Βιομηχανία, που είναι η υπεύθυνη για την ανακοίνωση όσον αφορά την ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Στηρίζουμε απόλυτα τις κατευθυντήριες γραμμές των προτάσεών μας. Υπάρχουν όμως δύο σημεία που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να θίξουμε εδώ. Για να δούμε τις επιπτώσεις που απορρέουν από τις προτάσεις σας. Που λαμβάνουμε υπόψη. Το έχει να κάνει με την παράγραφο 3. Βέβαια, δεν έχω δει τις συμβαστικές σας τροπολογίες Κοίταξα όμως κάποιες από τις αρχικές σας όπου μιλάτε για ένα δίκαιο καταμερισμό όσον αφορά τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν άνθρακα. Ενώ λοιπόν περιμένουμε βελτίωση όσον αφορά την απόδοση, για χαμηλό άνθρακα δηλαδή, από ολόκληρη τη βιομηχανία, οι επιχειρήσεις βιομηχανίε οι οποίε χρησιμοποιούν πολλή ενέργεια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την ευρωπαϊκή οικονομία. Άρα λοιπόν η αλλαγή αυτή είναι σαν να εννοεί μείωση στο μέγεθος της κατανάλωσης ενέργειας από τις επιχειρήσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό μήνυμα, αυτό που θα έπρεπε να στείλουμε. Επίσης, οι βιομηχανίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο αποδοτικές πολλές φορές από τις αντίστοιχες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρο εδώ τι ακριβώς εννοείται. Αν η απασχόληση περάσει από αυτές τις επιχειρήσεις, τις βιομηχανίες που καταναλώνουν πολύ ενέργεια και πάει σε άλλες που έχουν χαμηλότερο αποτύπωμα άθρακα, δεν είναι το σωστό μήνυμα πιστεύουμε εμείς. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως θα έπρεπε να ξαναδούμε τι θα κάνουμε με τον όρο shift στην πρόταση αυτή. Δεύτερον, πιστεύω ότι βάσει της δουλειάς που κάνουμε για τις τεχνολογίες και τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες για την ε, μικροηλεκτρονική, για παράδειγμα, και για άλλες τεχνολογίες. Εμείς ίσως εδώ θα έπρεπε να δούμε γενικότερα τις τεχνολογίες, όχι μόνο τις περιβαλλοντικές. Φυσικά και οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά υπάρχουν και άλλες που είναι επίσης σημαντικές. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είναι αναγκαίο να επιταχύνουμε τη δημιουργία μιας δικιάς μας αγοράς σε τέτοιες τεχνολογίες. Συγχρόνως πρέπει να αναλάβουμε δράση ώστε ο κόσμος να μπορεί να αναπτύξει τις δεξιοτεχνίες που χρειάζεται για να τις χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες ευρέως. Αυτά τα σχόλια είχα να κάνω. Κατά τα είπα, μας ικανοποιούν οι προτάσεις σας. Απλώς αναρωτιόμαστε για αυτά τα δύο σημεία μήπως θα έπρεπε να ξαναδούμε την ε, ισορροπία που πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει και την διατύπωση με τον όρο shift. Τις προτάσεις σας τις παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά και είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε την πλήρη διάσταση των προβλημάτων για τα οποία συζητάμε. Ωραία, ξαναρχίζει η συζήτηση για μας. Δεν ξέρω, εσείς θέλετε να αλλάξετε το shift κύριε Σιγητά. Μήπως θέλετε, πως έχετε κάποια άλλη αντίδραση, έχετε κάτι να πείτε. Ναι, βεβαίως ε, θα λάβουμε υπόψη αυτές τις απόψεις αλλά πιστεύω ότι η διαδικασία ήταν τόσο ταχεία που εγώ και οι σκιώδεις εισηγητές ε, συμφωνήσαμε σε αυτή τη λύση, αλλά φυσικά θα λάβουμε υπόψη και αυτές τις προτάσεις. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει συμφωνία ε, μεταξύ των ε, περισσότερων πολιτικών ομάδων για να προχωρήσουμε την πρόταση αυτή. Έτσι λοιπόν θα υιοθετήσουμε την παρατηρήσή σας. Μια που η ψηφοφορία για την γνωμοδότηση αυτή θα γίνει αύριο, υποθέτω ότι αν δεν ακούσουμε τίποτα άλλο, θα ψηφίσουμε το κείμενο που μας έχετε παρουσιάσει. Ήδη. Αυτό θα εξετάσουμε αύριο. Ωραία. Τώρα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Γιατί έχουμε κερδίσει χρόνο. Όλος παραδόξος. Η κυρία Καριμάντελή δεν είναι εδώ, δεν έχει έρθει. Ενώ είναι το δικό της σημείο που έχουμε τώρα να εξετάσουμε στην εμμυρίσια διάταξη. Οπότε, οπότε Διακόπτουμε για ένα τέταρτο της ώρας. Στις 5 και 25 να είσαστε εδώ. Συγγνώμη ζητάει από τους διερμηνείς οι Πρόεδρες και υπόσχεται να μην μας κρατήσει παραπάνω μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Bien, chers collègues, excusez-moi de cette méthode de travail qui n'est pas très agréable. Η μέθοδος αυτή εργασίας, λέει η Πρόεδρος, μπορεί να μην είναι ιδεώδης, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούσαμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες που έχουμε στην έκθεση της κυρίας Ντελή τη απουσία της. Τώρα λοιπόν που ήρθα μπορούμε να ξεκινήσουμε με το σημείο 7. Της δίνω λοιπόν και το λόγο για να εξετάσουμε τις 82 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στην γνωμοδότησή της που πάει στην Επιτροπή Πολιτισμού. Έχει να κάνει με την απελευθέρωση του δυναμικού του κλάδου πολιτισμού και δημιουργικότητας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που καθυστέρησα κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους και όδες εισηγητές και όλα τα μέλη της Επιτροπής μας που υπέβαλαν τόσες πολλές τροπολογίες που εμπλουτίζουν αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Αναγκαστήκαμε στο λίγο χρόνο που είχαμε στην διάθεσή μας να υποβάλουμε μόνο στα γαλλικά τις συμβαστικές ε, προτάσεις. Ευχαριστώ τους συναδέλφους πάντως για την κατανόηση που έχουν δείξει. Έχουμε 8 συμβιβαστικέ τροπολογίε λοιπόν που καλύπτει πάνω από τι μισέ τροπολογίε και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και τη Κομισιόν που θα φανεί και αύριο στην ψηφοφορία. Υπογραμμίζω τι διακυδεύεται και τι θελήσαμε να καλύψουμε με τις συμβαστικές μας τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να καλύψουμε το σημαντικό ρόλο που παίζει ο κλάδος στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά επίσης και προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους της στρατηγικής 2020 που είναι να βασιστούμε στη γνώση και στην κοινοτομία. Θέλω επίσης να αναφερθώ στις ιδιαιτερότητες των συνθηκών εργασίας του κλάδου αυτού. Ιδιαίτερα ό,τι έχει να κάνει με το ότι τα έσοδά τους παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν διακυμάνσεις και στα συστήματα κάλυψής τους για την περίθαλψη, την υγεία, την μητρότητα κλπ. Θέλουμε επίσης να βελτιώσουμε εδώ και ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση των νέων, με τη δημιουργικότητά του και να ενθαρρύνουμε την πρόσβαση των νέων στην απασχόληση σε αυτόν τον κλάδο. Όπως επίσης να μιλήσουμε και για την κινητικότητα και για την πολιτισμική ποικιλομορφία. Μιλάμε επίσης για την κατάρτιση, τη διαβίου κατάρτιση σε ένα κλάδο ο οποίο αλλάζει ταχύτατα. Έχουμε την ψηφιακή επανάσταση, έχουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επίσης του κλάδου αυτού που χρειάζονται στήριξη για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις μικροπιστώσεις, επί παραδείγματι. Επίσης, είμαστε θετικοί και απέναντι στις άλλες τροπολογίες που δεν καλύπτονται από τους συμβασμούς, αλλά που βελτιώνουν ουσιαστικά το αρχικό κείμενο, υπογραμμίζοντας το δυναμισμό που διαθέτει ο κλάδος υπέρ της ε, απασχόλησης. Ιδιαίτερα στηρίζω την τροπολογία 42 Κώστα Κοφεράτη για τι διαφορέ που υπάρχουν στου μισθού μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όσον αφορά τώρα τα πνευματικά δικαιώματα συγγραφέων εδώ και δημιουργών. Εδώ θεωρούμε ότι δεν είναι αρμοδιότητα τη δικιά μα επιτροπή, γι' αυτό και εδώ είπα ότι είμαι κατά των τροπολογιών 78 και 81. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη στάση, διότι θέλουμε σωστές αμοιβέ για ε, το δημιουργικό έργο. Όταν λέμε ότι πρέπει να ενισχύουμε όλο και περισσότερο τα πνευματικά δικαιώματα, προσοχή γιατί μπορεί να πετύχουμε το αντίθετο από αυτό που θέλουμε. Αντίθετα, εμεί θέλουμε περισσότερη απασχόληση, περισσότερη δημιουργία. Προσοχή λοιπόν στους κανόνες και στις εξαιρέσεις αυτό το τομέα. Είμαι στη διάθεσή σας για να σχολιάσω ό,τι θέλετε και όποια τροπολογία θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Στέλνουκ. Επιθυμώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια στο όνομα της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την θαυμάσια συνεργασία. Δεν έχω για την ώρα να συμπληρώσω τίποτε. Είναι σωστό που εκπονήσαμε την έκθεση αυτή ώστε να ευαισθητοποιηθούμε όλοι για ένα τομέα που δεν ε, βρίσκεται τόσο κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας και όμως αξίζει. Κύριος Μπαλτάσσαρ, ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση του ΕΛΚ για την ε, δραστηριότητα της ε, συντάκτριας. Ε, μπόρεσε να συμπεριλάβει τη συνεισφορά όλων σε συμβαστικές τροπολογίες και δείχνει πολύ μεγάλη ικανότητα σύνθεσης αλλά και τη δήλωση αυτής της Επιτροπής και την ικανότητά της να συγκλίνει επί των θεμελιωδών σημείων και η 38 ακόμη τροπολογίες που μένουν εκτός συμβαστικών προτάσεων είναι θετικές, επομένως εμείς θα ψηφίσουμε και υπέρ σχεδόν όλων των τροπολογιών. Υπάρχει σύγκληση λοιπόν επί των ουσιαστικών σημείων της έκθεσης. Το σημαντικό είναι ε, να δούμε πόσο προωθεί την ανάπτυξη ο τομέας αυτός για την Ένωση και πρέπει να προσδώσουμε ιδιαίτερη ε, σημασία στην ιδιαιτερότητα ε, τον ε, επαγγελματιών αυτών ε, και να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη δυνατότητα διεθνούς συνεργασίες. Έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι, εταιρείες, ε, οργανωτές και πρεσβευτές του πολιτισμού να κινηθούν σε μια πιο ευρία έννοια με σχέσεις με κρατη και με πρωτοβουλίες που να μεγεθύνουν τον τομέα αυτό και χρειάζεται φυσικά ε, και αναγκαιότητα να λάβουν ε, οι καλλιτέχνες καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτή είναι η άποψη και η δική μας. Είμαστε πολύ θετικοί απέναντι στην γνωμοδότηση και θα ήθελα και πάλι να αναφερθώ στο πόσο καλό έργο έκανε η συντάκτρια κυρία Ράπτη. και ευχαριστώ. Ορισμένα σχόλια από τον κύριο Στάρξ, ε, το σχεδίσει γιατί με ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την καλή δουλειά που έκανε και για την έκθεσή της. Ε, ο κ. Στάρξ είναι ικανοποιημένο με την κατεύθυνση που ακολουθεί αυτή η έκθεση. Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν μεγάλε δυσκολίε και λέει ότι μετά από διαπραγματεύσει με την εισηγήτρια οι φιλελεύθεροι μπορούν να υποστηρίξουν τι τροπολογίε. Μόνο ένα-δύο αιτήματα για την τροπολογία 12 που δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε, λέει η πρόσβαση στη γνώση και στο δημιουργικό πλαίσιο αποτελεί ε, μια ουσιαστική πτυχή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, και επίσης ε, θέλω να πιστήσω, θέλω με ένα σχόλιο από την συγκεκριμένη γι' αυτό και θέλω να πιστήσω την προσοχή σας και στο εξή για να μου πείτε πόσο σημαντικό είναι στη μόνη τροπολογία που έχω στα αγγλικά είναι η ΔΕΛΤΑ. D, γιατί στην αρχική παράγραφο 3 που έχει τροποποιηθεί χρησιμοποιήθηκε ο όρος residencies και στο συμβιβασμό λέγεται residences. Δεν είμαι σίγουρη γιατί ο όρος residency που τελειώνει σε Y έχει διαφορετική σημασία και νομίζω ότι πρέπει να διερευνήσετε τη διαφορά μεταξύ residency και residence. Και για την ε, τροπολογία 77 όπου μιλάμε για εγγύσεις, ε, για κεφαλαία εγγύσεων. Θέλω να ρωτήσω ποιος ε, είναι ο στόχος αυτών των εγγυητικών κεφαλαίων. Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε αυτό. Καταλαβαίνουμε τα φορολογικά κίνητρα, αλλά θέλω να μας ξεκαθαρίσετε το άλλο στοιχείο. Ευχαριστώ. Κύριε Änderungsantrag 77 Αποσύρεται η παριθμόν 77 τροπολογία, λέει η κυρία Στάινμπρουκ. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Ce n'est pas le cas. Madame Deli, vous avez la parole. Αν δεν ε, υπάρχουν εσπενεμβάσεις, κυρία Ντελή. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί αυτή, αυτό το έργο είναι και δικό μας έργο. Σας ευχαριστώ λοιπόν ειλικρινά που αφιερώσετε χρόνο να διαβάσετε το κείμενο και να ξέρετε αυτούς τους καλούς συμβιβασμούς, γιατί πραγματικά είναι προϊόν συλλογική ευφυία για την κυρία για την τροπολογία υπερθμών 12 που λέει ότι η πρόσβαση στη γνώση ε, και στο περιεχόμενο της δημιουργίας είναι στοιχείο θεμελιώδης γνώσης. Λέμε για την πρόσβαση στη γνώση εδώ, ότι η πρόσβαση στη γνώση είναι δικαίωμα Δηλαδή μιλάμε για τη γνώση, αλλά από τη σκοπιά της δυνατότητας της πρόσβασης. Και νομίζω όλοι έτσι το κατάλαβαν, εκτός από εσάς από τους φιλελευθέρους. Μήπως ε, ήταν πρόβλημα της μετάφρασης. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires Υπάρχουν άλλα σχόλια για τις ε, παρατηρήσεις της κυρίας Χαρκίνη για την παράγραφο 3. Εδώ, εδώ διαβάζω και τις δύο γαλλικές εκδοχές της ε, αρχικής παραγράφου 3 και της συμβιβαστικής. Βλέπω τον ίδιο όρο. Μιλάμε εδώ για χώρους κατοικίας και καλλιτεχνικά εργαστήρια. Δεν ξέρω στην αγγλική εκδοχή αν υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν έχει αλλάξει όρο στη γαλλική εκδοχή. και στις δύο περιπτώσεις λέγεται το ίδιο στο κείμενο. I'm just referring to Αναφέρουμε στην αρχική παράγραφο 3, στα αγγλικά. Η αρχική παράγραφος 3 τελειώνει σε λέει residencies, ISE, και στην τροπολογία λέει «residences» είναι διαφορετική η λέξη δηλαδή. Μπορεί να μην είναι σημαντικό, αλλά μάλλον υπάρχει απόκληση. Γιατί στα αγγλικά αναφερόμαστε σε έναν καλλιτέχνη ο οποίος ε, όταν είναι in residence σημαίνει ότι κάνει την πρακτική του. Σω κάποιο θα μπορούσε να μα ε, το ξεκαθαρίσει αυτό. Euh, euh, Τέλο πάντων έχουμε αυτή τη γλωσσική δυσκολία, αλλά κοιτάξτε η αρχική εκδοχή είναι η γαλλική εκδοχή. Έτσι λοιπόν αυτή είναι που ισχύει. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο για το κείμενο αυτό, θα ψηφίσουμε αύριο. Η Επιτροπή Επιτροπή, Επιτροπή Πολιτισμού θα ψηφίσει στις 25 Ιανουαρίου. Ας περάσουμε τώρα στα σημεία 8-13 της ημερής της διάταξης, όπου θα εξετάσουμε ένα πακέτο έξι κειμένων που αφορά την οικονομική διαχείριση, την οικονομική διακυβέρνηση. Έχουμε εδώ δύο εισηγητέ. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στον κύριο Δαβίτ Κάσα. Θα πρότεινα να παρουσιαστούν τα κείμενα το ένα μετά το άλλο και κατόπιν να οργανώσουμε την καθολική συζήτηση. Γιατί έχουμε πρώτη ανταλλαγή απόψεων εδώ, χωρί γραπτά κείμενα. Κύριε Σιγητά, για τα τρία πρώτα τροποποίηση του κανονισμού ε, για την επιτέχνηση και διασαφήνιση εφαρμογή διαδικασία υπερβολικού αγγλήματο. Το δεύτερο κείμενο έχει να κάνει με τι απαιτήσει για το δημοσιονομικό πλαίσιο των κρατών μελών. Και το τρίτο για ε, την εφαρμογή τη δημοσιονομική υποπτία στην Ευρωζώνη. Grazie signora Presidente. Um, Ευχαριστώ πολύ. Πέρασαμε από μια σημαντική κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πάρα πολλή δουλειά για να την αντιμετωπίσει και να αντιμετωπίσει κυρίως στις ευάλωτες περιπτώσεις. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική εποπτεία του οικονομικού τομέα, ούτε στα μάκρο, ούτε στα μικροοικονομικά συστήματα. Γι' αυτό θελήσαμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Όταν πρόκειται για τις αμοιβέ των δημοσιονομικό τομέα, επίσης προσπαθήσαμε να καθορίσουμε βασικές προδιαγραφές μέσω της τρίτης οδηγίας και εγκρίναμε κάποιους αυστηρούς κανόνες. Τώρα, Όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, βρισκόμαστε πίσω. Περιμένουμε η Επιτροπή να δημοσιεύσει τις έξι προτάσεις της που εμεί θα αναλύσουμε και θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες και εβδομάδες. Βλέπουμε πώς οι οικονομίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και πώς εφόσον υπάρχει αστάθεια στη μία χώρα, αυτή μετατοπίζεται και πηγαίνει και στις άλλες χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται πιο ξεκάθαρα όταν οι χώρες μέλη συμμετέχουν και στην Ευρωζώνη. Με μέτρα λοιπόν οικονομικής διακυβέρνησης θα μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα τα δημοσιονομικά των χωρών μελών και να εντοπίσουμε τις υπάρχουσες τάσεις, να δούμε κατά πόσο υπάρχουν ανισορροπίες μακροοικονομικά, αν υπάρχουν ε, προϋπολογισμοί στα κράτη-μέλη που δεν είναι ικανοποιητικοί και γενικότερα αν υπάρχουν κίνδυνοι ε, επειδή δεν ε, τηρούνται τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πάντως είναι ζωτική σημασία να έχουμε τους σωστούς μηχανισμούς στη διάθεσή μας και μάλιστα έγκαιρα. Μόνο έτσι θα μπορούμε να προλαμβάνουμε στο μέλλον κρίσης σαν ε, και αυτή ε, που ξεκίνησε πρόσφατα. Εμείς πρέπει να έχουμε ηγετικό ρόλο σε αυτά τα θέματα, διότι η απασχόληση είναι παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει λοιπόν όλοι οι παράγοντες που έχουν να κάνουν με την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις να λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια του θέματος που συζητάμε. Χρειαζόμαστε μια στέρεα βάση. Και αυτό θα το πετύχουμε εφόσον ε, έχουμε μια καλή γνωμοδότηση για την έκθεση πρωτοβουλίας που ετοιμάζει το Κοινοβούλιο. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, συμφωνούμε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει εποπτεία των πολιτικών απασχόλησης η οποία εποπτεί να λαμβάνει υπόψη και τις διασυνοριακές συνέπειες των εθνικών πολιτικών απασχόλησης. Δεύτερον, θα θέλαμε ενίσχυση της Επιτροπής Απασχόλησης. Τρίτον, είναι εσωτική σημασία οι εθνικοί προπολογισμοί να διαρθρώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζουν την ανάγκη για μακρόχρονο σχεδιασμό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική προστασία, η υγεία, τα συστήματα συνταξιοδότηση επίση και να ικανοποιούν όλου του πολίτε. Τέταρτο, θέλουμε κυρώσει οι οποίε μπορεί να χρειαστούν από παραβάσει στο σύμφωνο σταθερότητα να μην επηρεάζουν κονδύλια το οποίο είναι προς όφελος των ε, πολιτών. Οι στατιστικές επίσης πρέπει να είναι αξιόπιστες και να φροντίσουμε να συλλέγονται με αξιόπιστο τρόπο. Τώρα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα τα διατυπώσουμε όλα αυτά και να φροντίσουμε τα σημεία αυτά να συμπεριληφθούν στις τελικές εκθέσεις. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, σας παρουσίασα τις βασικές μου ιδέες για τα τρία αυτά θέματα. Εφεξής πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε τι ακριβώς θα προτείνουμε. Τέλος, θα συνεργαστώ με τους σκιώδεις εισηγητές και όλους τους συναδέλφους εδώ στην Επιτροπή αυτή για να καταλήξουμε στις καλύτερες δυνατόν λύσεις ώστε η τελική έκθεση να εγκριθεί όχι μόνο από την Επιτροπή μας, αλλά από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφε. Θέλω να παρουσιάσω και εγώ τα τρία, να πω τη γνώμη μου για τα τρία κείμενα. Και μετά θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της Επιτροπής που είναι εδώ εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης ΦΙΝ και που θέλουμε να μας εξηγήσουν λιγάκι τι θα γίνει και πώς θα λυθούν υπόψη οι δικές μας ανησυχίες. Ας ξεκινήσουμε με μια γενική παρατήρηση πριν μπω στην ουσία των τριών προτάσεων. Το πακέτο αυτό οικονομικής διακυβέρνησης, το είπε εξάλλου και υπουργό νωρίτερα, περιλαμβάνει πολλές πρωτοβουλίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με τις προτάσεις της Κομισιόν παρόλο που ξέρουμε ότι υπάρχει μια task force, μια ομάδα πίεση, η οποία, ε, μια task force, μια ομάδα τέλο η οποία ασχολείται και προσπαθεί να ε, συνεισφέρει, δίνοντας την άποψή της για τα έξι κείμενα που έχουν και τη σωστή νομοθετική μορφή. Αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση με το Συμβούλιο θα γίνει όταν θα έχει υιοθετήσει τη θέση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει, θα λάβει υπόψη και ό,τι γίνεται πιο πέρα. Αλλά δεν θα είναι αυτό που θα καθορίσει τη θέση του Κοινοβουλίου. Για τα τρία κείμενα λοιπόν που συζητάμε σήμερα και που πρέπει εγώ να σας παρουσιάσω. Θα αναφερθώ στο πρώτο. Έχει να κάνει με την ενίσχυση Ψάχνω να βρω τον τίτλο, λέει η κυρία Μπέρες. Πρόκειται για την ενίσχυση της εποπτείας και του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής. Πρόκειται για το σύμφωνο σταθερότητας. Πώς θα παληθεύουμε βάσει της εμπειρίας των τελευταίων δέκα ετών πώς θα μπορούμε να προλαμβάνουμε ε, κάποιες καταστάσεις και πώς θα αντιμετωπίζουμε τα υπερβολικά ελλείμματα των οικονομιών των χωρών μελών. Εκ μέρους της Επιτροπής μας λοιπόν δεν σκοπεύουμε να καλύψουμε όλο το θέμα, μόνο για την απασχόληση εμείς θα μιλήσουμε. Αλλά μετά από αυτά που ακούσαμε και από τον Υπουργό τελικά λαμβάνουμε υπόψη και τους άλλους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αποφασίσαμε με τη στρατηγική 2020. Θα ληφθούν υπόψη και αυτά τα στοιχεία. Και θα δούμε πώς την ανάλυση που θα κάνουμε θα πρέπει να δούμε και τα ελλείμματα αλλά και τα πλεονάσματα βάσει των κριτηρίων που θα έχουν αποφασιστεί στους δείκτες για τους οποίους θα σας μιλήσω σε λίγο. Όσον αφορά τώρα τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ξέρουμε ότι επηρεάζουν και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και τις συντάξεις και τον καθορισμό τους και γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων να συμμετέχει σε αυτόν τον μηχανισμό εποπτείας και να μην είναι μόνο το Συμβούλιο Κοφίλ που θα το κάνει. Για τα άλλα δύο κείμενά μου. Εκείνο για τα εκτελεστικά μέτρα όταν έχουμε υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες αλλά και όσον αφορά την διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών το ένα εξετάζει τις ανισορροπίες στο σύνολό τους και το δεύτερο μιλάει για μια πιο ειδική προσέγγιση όταν πρόκειται για τις χώρες της Ευρωζώνης. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Η πρώτη μου είναι η εξής. Πέρα από την μνήα στο άρθρο 121 πρέπει όπως είπαμε και νωρίτερα, να γίνεται μία και στο άρθρο 148. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι οι ανησυχίες μας όσον αφορά την απασχόληση αποτελούν μέρος της γενικότερης ανησυχίας για την μακροοικονομική ισορροπία. Αυτό πρέπει να φανεί από τον τρόπο με τον οποίο θα ετοιμαστούν οι διάφοροι δείκτες. Ακόμα και αν ε, δεν είναι η δικιά μας η Επιτροπή Αρμόδια για τα φορολογικά ζητήματα, παρόλα αυτά η ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών έχει σαν αποτέλεσμα το βάρος της φορολογίας σε σχέση με την απασχόληση επηρεάζει. Γι' αυτό πρέπει να δούμε και το φορολογικό. Έρχομαι τώρα στους δείκτες που για την πρώτη πρόταση είναι το κεντρικό στοιχείο. Γιατί από την ανάλυση των δικτών αυτών θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να προβλέψουμε μια κατάσταση ανισορροπίας συνολικά και να προβλέψουμε κυρώσεις. Το είπαμε ήδη. Εγώ όμως θα κάνω προτάσεις ώστε στο θέμα του ποσοστού απασχόληση ή το θέμα της ένδυα και του κοινωνικού αποκλεισμού να συζητηθούν και αυτά. Και να επαληθεύσουμε από τους διάφορους δίκτες να ληφθεί υπόψη αυτό που εμάς μας καίει. Είναι μια καινούρια στάση. Η πρόταση που μας έγινε για τον κανονισμό αυτό προβλέπει απλώς και μόνο ότι την αρμοδιότητα την έχει η Επιτροπή, η οποία αφού διαβουλευτεί με τα κράτη-μέλη θα συντάξει τους δείκτες. Μα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στον καθορισμό του πεδίου από το οποίο θα προκύψουν οι δείκτες. Τέλος και πάντα για τον εντοπισμό των ε, μακροοικονομικών ανισορροπιών, έχω να πω ότι σε αυτό το στάδιο ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Καμιά φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται. Αν χρειάζεται προπαρασκευαστική δράση. Όπως και με τις συστάσεις για τα μέτρα αυτά, το μόνο που γίνεται είναι ότι έρχονται και μας ενημερώνουν. Αλλά δεν γίνεται συζήτηση με το Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει σαφής μνήμα στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, ούτε γίνεται μνήμα στην διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τώρα το μηχανισμό κυρώσεων που προβλέπεται την περίπτωση μακροοικονομικών ανισορροπιών. Βάσει της διαπίστωσης λοιπόν ότι υπάρχουν μακροοικονομικές ανισορροπίες, η πρόταση που γίνεται είναι ότι σε περίπτωση υπερβολικών ανισορροπιών μέσα στην Ευρωζώνη, γιατί οι κυρώσεις αφορούν μόνο τα μέλη της Ευρωζώνης, προβλέπεται πρόστιμο. 0,1% μπορεί να φτάσει του ΑΕΠ της προηγούμενης χρονιάς για το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ο καρπός, δηλαδή τα χρήματα αυτά, μοιράζονται στις, στους καλούς μαθητές, στις χώρες που έχουν τηρήσει τις προδιαγραφές. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας προκυκλικός χαρακτήρας που δημιουργεί πρόβλημα όμως τι θα γίνει με τον ε, κοινωνικό προϋπολογισμό, τα κονδύλια, τα κοινωνικά και τι θα γίνει έτσι με την απασχόληση. Προτείνω λοιπόν να επανεισάγουμε κάποια στοιχεία ισορροπίας εδώ. Αυτά είχα να πω στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Αυτά έχω να σας προτείνω. Ακούσαμε και τον ε, David Κάζα. Πάντως, συνάδελφοι, αν συμφωνείτε, θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σερβαστερός, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής, αναπληρωτής γενικός διευθυντής στο ΚΦΙΝ, για να μας πει πώς αντιλαμβάνονται εκεί τις ανησυχίες της δικιάς μας Επιτροπής. Τι λένε, τι λέει το Συμβούλιο για τις ανησυχίες μας και τι περιθώριο βλέπετε εσείς να υπάρχει για συζήτηση μεταξύ μας. Και μετά θα συνεχίσουμε. Πριν να σας δώσω το λόγο, υπάρχει κάτι που εκπλήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τη σκοπιά της δημοσιονομικής διαδικασίας ε, επί της οποίας αναφέρθηκε ο Ντεβιτ Κάσα ε, υπάρχουν πολλές σκέψεις σε σχέση με το περιεχόμενο και όμως δεν υπάρχει τίποτα για το χρονοδιάγραμμα. Βλέπουμε ότι υπήρχε μια σχεδόν διακυβερνητική συμφωνία για ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο που όμως δεν αναφέρεται καθόλου στο κείμενο, δεν μεταφράζεται στο κείμενο, είναι εκούσιο αυτό. Υπάρχει κάποιος λόγος ενωτέρας βίας που δεν αναφέρεται υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Ε, δηλαδή έχουμε ένα πακέτο εξεκειμένων που είναι στη συναπόφαση και έχουμε και κάτι που δεν ξέρουμε το οποίο, το οποίο θα καταλήξει πού και πώς. Good evening, uh, Chair. Thank Καλησπέρα σας, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφράσουμε τις απόψεις μας για το ζήτημα. Ζητώ συγγνώμη που ξεκινήσα, που, συγγνώμη, που ήρθα καθυστερημένος και δεν μπόρεσα να ακούσετε δύο πρώτα λεπτά της παρουσίασης του κυρίου Κάζα, αλλά θα συζητήσουμε διμερώς. Και φυσικά ευχαρίστως να συζητήσουμε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να θέσετε σε σχέση με τα έγγραφα που παρουσίασε η Κομισιόν. Θα είμαι σύντομο, έτσι ώστε να σας δώσω και χρόνο για τη συζήτηση. Καταρχήν, ε, να τονίσω, όπως είπατε και στην παρουσίασή σας, ε, Πρόεδρε, ότι το πακέτο τη Κομισιόν, που παρουσιάστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, ε, είναι στο κέντρο της συζήτησης και οι συζητήσεις και με και με το Συμβούλιο προχωρούν. Υπήρξε μια παράλληλη διαδικασία ε, μέσω της Tax Force του Φανερομπόη, αλλά τώρα ε, έχουν φτάσει τα έγγραφα αυτά ε, στις ομάδες του Συμβουλίου και θα συζητηθούν και τα κείμενα της Κομισιόν. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά από την Task Force υπό την καθοδήγηση του Πρόεδρου Φανερομπόη, αλλά τώρα θα πρέπει να διοχετευτεί το έργο στα κανονικά βήματα, δηλαδή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του πακέτου της Κομισιόν της 29 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το θέμα αυτό και αν υπήρξε κάποιο δισταγμό ή αμφιβολία, ελπίζω να τη διασκέδασα πλήρω. Ε, τώρα, να μπούμε πολύ γρήγορα στην ουσία, αλλά να τονίσω καταρχήν πόσο σημαντική είναι η συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο και με τη δική σα Επιτροπή, αλλά και με άλλε επιτροπές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά πολύ καθοριστικές ε, στιγμές ε, για τον καθορισμό της Ευρωζώνης ε, και αυτές τις μέρες οι αγορές στέλνουν πολύ ηχηρά μηνύματα και αμφισβητούν την ικανότητα της Ένωσης να αναλάβει δράση. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και μέσω αυτής της δουλειά που κάνουμε να βελτιώσουμε την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει την ικανότητά της να δράσει τολμηρά και ταχαίως σε κάποια ζητήματα ζωτικά. Το δεύτερο εισαγωγικό στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι ενθαρρυνθήκαμε από τις διάφορες συζητήσει ε, που υλοποιήσαμε με ε, πολλούς από εσά ε, και άλλοι συναδελφοί μου από την Κομισιόν. Είχαν συζητήσεις με, άλλους, με άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όσα ακούσαμε μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά και ελπίζουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, επί της ουσίας είναι σαφές ότι αυτό το πακέτο που υιοθέτησε η Κομισιόν έχει ως βασικό στόχο να απαντήσει στα σύντομα σχόλια και δυναμίες ε, των ε, ε, δομών διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Τα κύρια προβλήματα είναι οι οικονομικές και χρηματοπιστικές ανισορροπίες και ε, στοχεύουμε στο να αποφύγουμε τέτοιες οικονομικές κρίσεις που βιώνουμε αυτές τις μέρες και ήδη αρκετό και, εδώ και κάποιο καιρό. Έτσι λοιπόν το πακέτο ε, δεν στοχεύει σε όλο τον κύκλο αλλά σε ένα τμήμα. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν αποφάσισε να προωθήσει κάποιες ανακοινώσεις για να αντιμετωπίσει τρία κυρία ζητήματα. Το ένα είναι το φορολογικό που θέλουμε να ενισχύσουμε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης με διάφορες προτάσεις. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες, ε, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Τα έχετε στη διάθεσή σας τα κείμενα. Το σημαντικό εδώ είναι να τονίσουμε ότι πρέπει να ε, τονίσουμε, να ενισχύσουμε το σκέλος της πρόληψης, αλλά θα πρέπει ε, να επικεντρωθούμε και επί της ουσίας. Έχουμε δύο πακέτα, δύο στοιχεία έχουν ισχυθεί το δημοσιονομικό πλαίσιο και ο εισηγητής εργάζεται από αυτού και αυτό είναι ένα από τα κύρια στοιχεία που έλειπαν στις δομές διακυβέρνησης μέχρι τώρα. Έτσι λοιπόν το να έχουμε εθνικά δημοσιονομικά ε, πλαίσια που επαληθεύουν αυτό που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι σημαντικό προκειμένου να έχουμε κυριότητα των δημοσιονομικών κανόνων που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουμε ε, να υπάρχει ίδια κυριότητα και σε εθνικό επίπεδο ε, και συζητήθηκε στο Συμβούλιο γιατί χρειαζόμαστε μια οδηγία. Ε, γι' αυτό πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια οδηγία. Τα περισσότερα κράτη-μέλη είναι υπέρ μια οδηγία γιατί βοηθά τα κράτη-μέλη να επανεισάγουν σε εθνικό επίπεδο τους δημοσιονομικούς κανόνες και πλαίσια που χρειάζονται και φυσικά οι χώρες αυτές με επικεντρωμένα ε, συστήματα είναι πολύ σημαντικό για αυτές να έχουν μια οδηγία που θα τις βοηθά να ε, επανισάγουν ε, αυτού του είδους το πλαίσιο με κατάλληλο τρόπο στις περιφερειές τους. Έτσι λοιπόν, πολλά κράτη-μέλη υποστηρίζουν την ύπαρξη οδηγίας. Ορισμένοι δεν έχουν πιστεί ακόμα, αλλά αυτή είναι η συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Και πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη οδηγία. Κατόπιν έχουμε τους μηχανισμούς επιβολής, συζητήθηκαν επί μακρόν. Εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ε, θέλουμε να έχουμε έναν αυτόματο χαρακτήρα, αλλά όχι απόλυτα αυτόματο χαρακτήρα, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη μέσω αυτής της αντίστροφης ε, πλειοψηφία ε, να γνωστοποιήσουν τις θέσεις τους αν υπάρχει λόγος. Ένα τμήμα για τις ε, κυρώσεις πρέπει να πτυχθεί περαιτέρω, έχουμε ένα σύστημα κυρώσεων για τις κυρώσεις, για το HDP και πρέπει να συζητήσουμε ακόμη τις κυρώσεις που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσω ενός γενικού νόμου, αλλά πρέπει να εισαχθούν διάφοροι μηχανισμοί κυρώσεων μέσω διάφορων κανονισμών που ε, θα διέπουν το θέμα αυτό και ε, άκουσα τι είπε ο πρώτος για το θέμα αυτό Πρέπει να τονίσουμε ότι οι κυρώσεις ε, δεν ε, θα επιβάλλονται κατά μεμονωμένων πολιτών, ε, θα επιβάλλονται σε εθνικό επίπεδο οι κυρώσεις. Δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τι ιδιωτικέ πρωτοβουλίε ή την ιδιωτική ανάληψη πρωτοβουλία. Και κάτι ακόμη, το θέμα των ανισορροπιών. Συζητήθηκε πολύ το ζήτημα αυτό, είναι κάτι καινούριο και πρέπει να το δούμε μαζί με ε, το με ένα ακόμα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε, το scoreboard. Αυτό το βαθμολόγιο πρέπει να το συζητήσουμε και από κοινού. Πρέπει να δούμε ποιος είναι ο στόχος του βαθμολογίου και πώς θα εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν θέλω να τονίσω ότι το scoreboard, αυτό το βαθμολόγιο θα έχει 8 με 10 δείκτες, είναι ακόμα υποκατάρτιση, υποεκπώνηση, δεν ε, έχουμε φτάσει ε, σε ολοκληρωτική εκδοχή, συζητούμε ακόμα με τα κράτη-μέλη και σίγουρα θα ζητήσουμε ένα περιορισμένο αριθμό δικτών, 8 με 10 δεν θέλουμε να έχουμε ένα ευρύ σύνολο γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε ιδιαίτερα πολύπλοκο εργαλείο στη συνέχεια. Ε, έτσι λοιπόν το scoreboard θα πρέπει να δοθεί ως ένα φίλτρο μέσω του οποίου θα εκτιμούμε σε ένα πρώτο επίπεδο την κατάσταση στα κράτη-μέλη και θα βλέπουμε σε ποιο επίπεδο φτάνουν οι ισορροπίες. Θα έχουμε κατόφλια, μέγιστο κεμά και θα έχουμε ε, κατόφλι και ανώτατο όριο ε, και κατόπιν ε, θα έχουμε διάφορα χρώματα σε αυτό το βαθμολόγιο. Ε, θα είναι πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο, αναλόγως με το βαθμό της σοβαρότητας της ανισορροπίας και κατόπιν θα προβαίνουμε σε ένα δεύτερο που θα είναι μια εις βάθος αναθεώρηση όμως το Σκολμπόρτ απλώς είναι ένα εργαλείο φιλτραρίσματος για να δούμε ποια είναι τα κράτη-μέλη που μπορεί να έχουν ε, πιθανότατα ανισορροπίες και να έχουν προβλήματα και ποια δεν έχουν και θα συζητηθεί φυσικά αυτό το θέμα με το Συμβούλιο του Σκορμπόρτ, αλλά εδώ θέλω να σας πω ότι η Κομισιόν θα έχει πλήρες δικαίωμα πρωτοβουλία για το δεύτερο βήμα, για να υπάρχει βάθο αξιολόγηση της ε, ενδιαφερόμενης χώρας. Αυτό δεν θα ε, εξαρτάται από το Συμβούλιο. Φυσικά θα ακούσουμε τις απόψεις ε, του Συμβουλίου και θα εμπλέκεται και το Κοινοβουλίο στο εγχείρημα, αλλά η Κομισιόν θα αναλάβει την πρωτοβουλία Και φυσικά αυτό θα γίνει και σε συνεργασία με τους ε, άλλους πρωταγωνιστές. Τώρα, ο ρόλος του Κοινοβουλίου στο βαθμολόγιο, στο scoreboard. Όπως θα δείτε, προτείναμε να έχουμε αναθεώρηση του scoreboard σε τακτική βάση κάθε τρία χρόνια, ε, γιατί το πράττουμε αυτό γιατί κάθε κρίση είναι διαφορετική εκφύσεως, το γνωρίζετε. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε πολύ καθορισμένο βαθμολόγιο που απαντά στη σημερινή κρίση, μπορεί να μην μπορεί να απαντήσει στην επόμενη κρίση. Έτσι λοιπόν, η ιδέα είναι να δοκιμάζεται αυτό το scoreboard ε, και να χρησιμοποιείτε τις σία καθώ θα εξελίσσεται η οικονομία και θα βλέπουμε νέα χαρακτηριστικά και θα τροποποιείται ε, αυτό το βαθμολόγιο και φυσικά θα συμμετέχουν και διάφοροι ενδιαφερόμενοι. Έτσι λοιπόν δεν θέλαμε να έχουμε κάτι σταθερό για πάντα αλλά κάτι υπό εξέλιξη προκειμένου να μπορούμε να αντικατοπτρίζουμε και τις διάφορες οικονομικές εξελίξεις και να είμαστε σίγουροι ότι ε, δεν θα ε, μας ξεφύγουν οι μελλοντικές ανισορροπίες και δεν θα έχουμε αποτυχία του συστήματος. Ε, δεν έχουμε πρόβλημα να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είδαμε ότι και στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχουν αποκλίνουσε απόψει σε σχέση με το βάθμο εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαρίστω ε, να συζητήσω και το, με το Συμβούλιο, Πρόεδρε, αλλά από ό,τι κατάλαβα, κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα, θέλ, θα ήθελαν ε, να βασιστούν στο 290 τις συνθήκες, τις για να ε, σχηματίσουν ε, μια ομάδα που θα συζητήσει το θέμα αυτό, ενώ άλλοι δεν θεωρούν ότι είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Εμείς κατανοούμε και το έχουμε συζητήσει με τον Επίτροπο άτυπα ότι το να δημιουργηθεί μια αντιπροσωπεία ίσως ε, θα είναι υπερβολικό, υπερβολικά επαχθές αλλά το συζητούμε το πώς θα μπορούσε το Κοινοβουλίο να δραματίσει το ρόλο που του αρμόζει ενώ θα διατηρούμε και ευέλικτη τη διαδικασία. Ένα άλλο θέμα είναι ο συνδέσμος με την ανάπτυξη αυτό που παρουσιάσαμε στο πακέτο αυτό είναι μόνο ένα τμήμα ε, των ε, ζητημάτων διακυβέρνησης ή διαχείρισης αν θέλετε αλλά θα έχουμε και άλλες προτάσεις στο μέλλον δεν εφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα παρουσιαστεί από την Κομισιόν ε, μάλλον παρουσιάστηκε τον Ιούνιο από την Κομισιόν και τώρα συζητείται και θα εφαρμοστεί για το 2011 εδώ τώρα η Κομισιόν θα παρουσιάσει την ετήσια ε, μελέτη για την ανάπτυξη, Annual Growth Survey, η ιδέα είναι να παρουσιαστεί νωρί τη διαδικασία και να δώσει κάποιους γενικούς προσανατολισμούς στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το σχεδιασμό πολιτικής για το 2011 και 2012. Δεν πρόκειται για μεσοπρόθεσμη στρατηγική, αλλά αυτή η Annual Growth Survey θα στοχεύει βραχυπρόθεσμα στο 2011 και στο 2012 και θα λαμβάνονται υπόψη και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα προγράμματα σταθερότητας και συγκλήσεις που θα παρουσιάσουν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα παρουσιάσουν ε, νέα τέτοια προγράμματα το αργότερο μέχρι τα μέσα ή τέλη Απριλίου, το αργότερο. Και αυτό θα επιτρέψει στην Κομισιόν να αξιολογήσει τα προγράμματα αυτά και στη συνέχεια να παρουσιάσει ολοκληρωμένες συστάσεις μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Αυτή είναι η διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Ξάμεινο. Ε, πρώτη φορά θα εφαρμοστεί. Ε, δεν ε, μάλλον θα έχουμε μια πιλωτική αν θέλετε εφαρμογή, δηλαδή θα ε, πράττουμε και θα μαθαίνουμε από αυτό. Έτσι λοιπόν, ε, το ευρωπαϊκό εξάμεινο που θα ξεκινήσει από το χρόνο θα είναι πολύ χρήσιμο. Τώρα, το δεύτερο ε, σύνολο κειμένου που έχει εγκριθεί έχει, να, έχει προκύψει από συνεργασία σε πρώτη ανάγνωση ε, και πρόκειται για για το Stability Board θα ξεκινήσει το πρώτο εγχείρημα τον Ιανουάριο. Επίσης, το Μάιο θα έχουμε δύο νέους ε, μηχανισμούς χρηματοδοτικούς. Ε, πρόκειται για άλλους δύο μηχανισμούς που θα μεταρρυθμιστούν στο μέλλον, θα μεταμορφωθούν στο μέλλον και θα δημιουργήσουμε δύο μόνιμους μηχανισμούς σταθερότητας. Έχουν συζητηθεί ήδη μια σειρά αρχών και έχουν δημοσιευτεί. Έτσι λοιπόν συνεχίσετε το έργο μας και για αυτούς τους μόνιμους μηχανισμούς σταθερότητας εν ώψη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου. Και το τελευταίο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδέεται πολύ στενά με το έργο σας εδώ. Πρόκειται στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 που έχει δημοσιεύσει η Κομισιόν θα ξεκινήσει το, ξεκίνησε το Μάρτιο φέτος. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Μέσο για την πρόθεση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί το κύριο μέσο που ε, αναπτύσσουμε τώρα και ε, συνδέεται πάρα πολύ στενά με όσα συζητάμε εδώ με την δομή διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε τη στρατηγική του 2020 να την συνδέσουμε με το πακέτο της 29 η ε, Σεπτεμβρίου. Το πακέτο αυτό ε, επικεντρώνεται στις μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες και στις δημοσιονομικές ανισορροπίες, όμως είναι σαφές ότι θα πρέπει να έχουμε μια στασμένη διαχείριση και των στοιχείων αυτών και δεν θα πρέπει να έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο όπου θα βάλουμε τα πάντα, δεν θα ήταν ε, καλό κάτι τέτοιο. Δεν λέω ότι ζητάτε κάτι τέτοιο πρόεδρε, ε, απλώς ε, καμιά φορά από αυτά που ακούμε έχουμε την εντύπωση ότι κάποιοι θέλουν όλοι στο όχι τη στρατηγική του 2020 να μπουν στο πακέτο της διακυβέρνησης και εμείς δεν θεωρούμε ότι θα βοηθούσε κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στο δημοσιονομικό σκέλος Όσο ε, μεγαλύτερη η σταθερότητα δημοσιονομική έχουμε, τόσο το καλύτερο βλέπετε ότι κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης αυτή η αστάθεια μας οδήγησε σε καταστροφικές συνέπειες ε, και στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από τη θεραπεία και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με αυτό το πακέτο της 29 η Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Euh, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας θα δώσω λόγο στους συναδέλφους. Πρώτα η κυρία Τουρούνιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω δανέζικα τώρα. Πρώτα θα ήθελα να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ταχύτητα σύνθεσης μιας αντιπροσωπείας δεν είναι πρόβλημα για μας. Μπορούμε να την φτιάξουμε γρήγορα, αν θεωρείτε ότι είναι πρόβλημα αυτό. Τώρα, για τα έξι αυτά σημεία. Μόλις κάναμε μια κοινή συζήτηση για αυτά τα έξι θέματα. Αλλά θα έπρεπε να, τα έχουμε, να έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια το θέρος του 2011. Αλλά βλέπουμε τους κινδύνους ότι δηλαδή οι εξελίξεις μας ξεπερνούν. Βλέπε το παράδειγμα της Ιρλανδίας γιατί οι κερδοσκόποι συνεχίζουν και μετά θα επιτεθούν στην επόμενη χώρα και στην μεθεπόμενη. Υπάρχει λοιπόν μια εξελισσόμενη κατάσταση ιδιαίτερα δραματική και ανάμεσα στις φάσεις αυτές της ε, ε κατάστασης προσπαθούμε να περάσουμε κάποιες νομικές διατάξεις που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο ενώ ταυτόχρονα ολόκληρο το σύστημά μας ε, ε, διακινδυνεύει, βρίσκεται σε κίνδυνο μάλλον. Αλλά πρέπει να κάνουμε δουλειά αυτή. Τώρα για μας τους πράσινους. Αυτό που θεωρούμε εμεί ότι είναι σημαντικό σχετικά με τις νέες νομοθετικές ιδέες πρέπει να είναι ο στόχος. Όσο να αφορά το στόχο θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση μιας στέρεας υγιούς οικονομίας. Όχι μόνο των ε, δημόσιων οικονομικών, αλλά σε όλο τη το φάσμα. Δεύτερο, ενίσχυση της απασχόλησης. Τρίτο, μια βιώσιμη οικονομία. Τέταρτο, να υπάρχουν και σωστές, να εξασφαλίζονται σωστές δομές διαχείρισης, governance, τη κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει όμως αλλαγές. Συμφωνούμε, έτσι το βλέπουμε και εμείς. Χρειάζονται λοιπόν σημαντικές αλλαγές στο μέχρι τώρα σύστημα, όσο εδώ καλά. Αυτό τώρα όμως που προτάθηκε από την Κομισιόν στις 29 Ενάτου, χρειάζεται ακόμα πολλές βελτιώσεις, έτσι το βλέπουμε εμείς τουλάχιστον. Θα έρθω σε ορισμένα σημεία τώρα που για μας έχουν κέριο χαρακτήρα. Πρώτο, η ταχύτητα, ο ρυθμός. Πρόκειται για τον ρυθμό της μείωσης του χρέους και του ελλείμματος. Είναι σημαντικό. Να είναι σωστός ο ρυθμός, να είναι επαρκής ο ρυθμός, να μην δυσμονούμε όμως τις κοινωνικές επιπτώσεις. μείωση των χρεών κατά το 1 εικοστό ανά έτος, να δούμε ε, αν ο ρυθμός αυξηθεί στην μείωση του χρέους και του ελλείμματος. Και βέβαια πρέπει να αποδομηθούν το χρέος και το έλλειμμα, αλλά πόσο γρήγορα και τι γίνεται με τις κοινωνικές επιπτώσεις. Δεύτερο, οι ε, κυρώσεις, θέματα 10 και 11 στην ημερήσια διαταξή μας. Όπως είπε και η Πρόεδρος, Μπορεί να είναι κανείς προκυκλικός. Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο κυρώσεις, όχι μόνο δηλαδή το καμτσίκι, αλλά και η επιβράβευση, η ζάχαρη. <clears throat> Χρειάζεται μια συνολική αξιολόγηση της οικονομίας μιας χώρας που πρέπει να γίνει πριν να επιβληθούν κυρώσεις. Οι κυρώσεις δηλαδή δεν μπορούν να επιβάλλονται αυτομάτως. Επίσης τώρα για τις κυρώσεις έχω μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Ακούστηκαν πολλά σχετικά με την επέκταση των κυρώσεων και επιβολή σε χώρες μη ζώνης ευρώ μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού με ανακοπή με αναστολή πληρωμής πιστώσεων για παράδειγμα από τον αγροτικό προϋπολογισμό. Τώρα, οι μακροοικονομικοί δείκτες θα είναι πολύ σημαντικό πώς θα διαμορφωθούν. Και είναι σημαντικό εδώ να μπορεί να συμμετάσχει το Κοινοβούλιο. Η αντιπροσωπεία, την αντιπροσωπεία τη φτιάξουμε. Πάντως, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ακριβής διαμόρφωση του βαθμολογίου. Είναι σημαντική. Είναι σημαντικό και να συζητήσουμε τι σημαίνει δηλαδή τώρα για την Ευρώπη ότι η Γερμανία έχει αυτή την οικονομική ανάπτυξη. Έχει αυτό το μοντέλο εξαγωγών. Γίνεται στην πλάτη των υπολείπων της Ευρώπης και τι θα γίνει εάν εξοικονομεί ολόκληρη Ευρώπη. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ των χωρών μελών της Ευρώπης. Επίσης, δεν είναι δυνατό η οικονομική πολιτική όλων των χωρών μελών να εναρμονιστεί, να γίνει ενιαία. Χρειάζεται μια ανοιχτή συζήτηση για τον εσωτερικό δυναμισμό και τις εσωτερικές διασυνδέσεις. Εάν λοιπόν το βαθμολόγιο γίνει σωστά, πρέπει να γίνει. Αλλιώς ε, το όλο αυτό θα καταλήξει να είναι μια φάρσα. Ολοκληρώνοντας, έχω να πω το εξή. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να τροποποιηθεί σε ορισμένα σημεία, ώστε να επιτρέψει μια κατεύθυνση της οικονομίας με ε, κοινωνική ευθύνη. Η κυρία Χάρκιν, ως και ο συγκητής μας ε, κολλείεται δυστυχώς σε χωρισμένα σχόλιά του, αλλά σημειώνω ότι δεν συμφωνώ με τα σχόλια αυτά, όμως με παρακάλεσε να τα διαβάσω. Λέει ότι συμφωνεί με την νομοθετική πρόταση για την οικονομική διακυβέρνηση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν ισχυρό ε, ε, κοινοτικό προϋπολογισμό και μια σταθερή οικονομική ανάπτυξη που θα διατηρήσει την απασχόληση. Πιστεύει ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κανονισμό θα πρέπει να διαμορφωθεί με πολύ πιο αποτελεσματικό και υποχρεωτικό τρόπο η αντίστροφη πλειοψηφία του Συμβουλίου είναι σωστή όταν αναφέρεται στην λήψη κυρώσεων, στην επιβολή κυρώσεων μάλλον σε μια χώρα μέλος. Πρέπει όμως να είναι ακόμα σοβαρότερες οι επιπτώσεις εάν μια χώρα αποδεικνύεται ότι δεν διαθέτει δημοσιονομική πειθαρχία. Χρειαζόμαστε και νέες κυρώσεις από το λεγόμενο naming and shaming μέχρι το προσωρινό πάγωμα ευρωπαϊκών πόρων μέχρι την οριστική απώλεια ευρωπαϊκών πόρων και την επιβολή οικονομικών ε, κυρώσεων. Δεύτερο, συνεχίζει ο σκέδιος χρειαζόμαστε ένα πλήρως αυτοποιημένο μηχανισμό κυρώσεων, όπου δεν θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι χώρες ε, μέλη. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία των χωρών μελών και να αποφύγουμε νέα προβλήματα όπως αυτά της Ελλάδας και της Ιρλανδίας που επιβαρύνουν τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Βρίσκω δύσκολο να διαβάσω την τελευταία του πρόταση, αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσω γενικά μου θα κάνω ένα σχόλιο και μετά θα έρθω στα δικά μου σχόλια να τα βάλω τα πράγματα αυτά σε κάποιο πλαίσιο. Τα προβλήματα της Ελλάδος και της Ιρλανδίας είναι πολύ διαφορετικά και τα δύο είναι πολύ σοβαρά και βεβαίως έχουν ευθύνη και οι δύο χώρες αλλά τα θέματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Ασφαλώς στην Ιρλανδία αυτό που συνέβη είναι επειδή τα πιστοτικά ιδρύματα στην Ευρώπη ολόκληρη επένδυσαν χωρίς κανένα, ε, καμιά αναστολή στα τραπεζικά ιδρύματα της Ιρλανδίας. Πάλι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Βλέπε Πορτογαλία και Ισπανία και δεν ε, λύγει ο κατάλογος εκεί. Και γίνονται όλο και πιο τρομακτικά τα πράγματα. Εάν ακούσουμε τώρα ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες, παράδειγμα η καγκελάριος Μέρκελ, έχει μια τελείως διαφορετική οπτική για όλα αυτά θα πληρώσουν αυτοί που φταίνε. Αλλά για την ώρα οι φορολογούμενοι πληρώνουν το λογαριασμό. Κάνω το γενικό σχόλιο. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κοινό στόχο σε ό,τι με αφορά. Τώρα ο κύριος Κάζα, ή μάλλον κύριε Κάζα, ίσως να μην καλά τη μετάφραση. Ε, είπατε η κρίση που περάσαμε. Εγώ λέω η κρίση που περνούμε ακόμα μιλήσατε για το ότι οι αγορές αμφισβητούν την ικανότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλούμε για το μέλλον, μιλούμε όμως και για το παρόν που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Και ασφαλώς για το μέλλον χρειαζόμαστε σχεδιασμό. Μία ερώτηση προς την Κομισιόν είναι η εξής. Οι προτάσεις που ε, κατατίθεται θα σημάνουν αναθεώρηση της συνθήκης και σε ποιο επίπεδο. Και κυρίως όταν μιλάτε για την λεγόμενη reverse majority αντίστροφη πλειοψηφία και άλλα θέματα. Δεν έχω διαβάσει τα έγγραφα, το ομολογώ. Έριξα μια ματιά σε ορισμένα, αλλά δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα. Έχω διαβάσει άλλα βέβαια. Μέχρι την επόμενη συζήτηση όμως θα τα έχω διαβάσει. Μπορώ να θέσω ένα άλλο ερώτημα πριν να έρθω σε ορισμένα από τα ειδικότερα θέματα και δεν θα μακρηγορήσω. Όλοι κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τον ελέφαντα μέσα στο, στην αίθουσα που είναι το ερώτημα το, η αρχιτεκτονική που έχουμε για την υποστήριξη του κοινού νομίσματος είναι επαρκής. Χρειαζόμαστε μεταφορές από την Ένωση για να, επι, δηλαδή, για να επιβιώνει το ευρώ. Καλές ιδέες για την καλή διαχείριση, αλλά θα είναι επαρκές για τη στήριξη του νομίσματος μέσω και μακροπρόθεσμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΕΠΣΚΟ και μίλησε ο κ. Κάζα προηγουμένως και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η κυρώσει δεν θα πλήξουν του πολίτε. Μίλησε για παράδειγμα για τα συνταξιοδοτικά ε, συστήματα. Θα είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε αυτό και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στα πλαίσια της δικής μας εδώ της Επιτροπής για να διασφαλίσουμε αυτή την ε, ορθή έκφαση. Αλλά σε τελική ανάλυση, ανεξαρτήτως του τι θα πράξουμε, οι κυρώσεις θα πλήξουν τους πολίτες με κάποιον τρόπο. Και ακόμα και αν δεν μιλούμε πολύ για την Ιρλανδία, μας πήραν το μισό συνταξιοδοτικό σύστημα για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Εάν λοιπόν μπορώ να κρίνω από τα πράγματα που συμβαίνουν σήμερα, οι, ε, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι βαριές για τους ε, πολίτες. Η κυρία Τούρουνεν μίλησε προηγουμένως για την ανάγκη τήρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και για τις επιπτώσεις. Δεν θα πω περισσότερα, το εξήγησε η ίδια πάλι για τις κυρώσεις. Συμφωνώ με την κυρία Μπερές όταν λέει για τα πρόστιμα που θα πάνε από τις κακές εντός εισαγωγικών χώρες μέλη τις καλές με αυτή, αυτό το προκυκλικό χαρακτήρα. Αλλά θα τα δεχθούν αυτά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και τέλος, πάλι για το βαθμολόγιο. Επαναλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω αρκετά, γι' αυτό κάνω μια ερώτηση επειδή είναι διαφορετικά διαθρωμένες οι οικονομίες μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες έχουν πλεόνασμα, άλλες έχουν έλλειμμα, το βαθμολόγιο πώς θα τα πάρει υπόψη του όλα αυτά τα πράγματα και θα μας προσφέρει την ανάλυση που χρειαζόμαστε. Δύο λεπτά έχουμε ακόμα με τους ε, διερμηνείς, γιατί έχω ήδη υποσχεθεί ότι θα τους αφήσουμε να φύγουν ε, στην ώρα τους. Εάν οι συνάδελφοί μου θέλουν να συνεχίσουμε τη συζήτηση, θα το κάνουμε στα αγγλικά, αλλά θέλετε να... Κύριε Χέντερ, θέλετε να παρέμβετε. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις τους στους συναδέλφους. Είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να μπορέσει να τοποθετηθεί, γιατί στην κλίμακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχουμε άλλη δυνατότητα προσέγγισης και να απαντήσουμε στις ανησυχίες των αγορών. Γι' αυτό το λεγόμενο μείγμα πολιτικής δημιουργίας απασχόλησης και το ρόλο που έχει απασχόληση για την αποκατάσταση των δημοσίων οικονομικών. Αν επιτρέπετε κύριε Ντερόζ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια ερώτηση που μπορείτε να απαντήσετε στα αγγλικά και έτσι μπορούν να αποχωρήσουν οι διερμηνήσεις όταν θα τελειώσουμε αυτή. Πού βρίσκονται οι συζητήσει αυτή τη στιγμή στου κόλπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά μια ενδεχόμενη αναθεώρηση των συνθήκων. Διότι είδαμε ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι τέθηκε επιτάπητος ε, το σενάριο αυτό. Και νομίζω ότι όσο μιλάμε κρυμμένα, τόσο το καλύτερο, έτσι πιστεύουν ορισμένοι. Εάν θεωρήσουμε ότι πρέπει να ξανανοίξει η συνθήκη της Λισαβόνας για την οικονομική διαχείριση μόνο για να συζητηθεί το θέμα που προβλέπουν θα ήταν πάρα πολύ αντιπαραγωγικό το μήνυμα αυτό ακριβώς όπως λέει και η κυρία Χάρκιν δηλαδή Θέλουμε να προχωρήσουμε στην οικονομική διαχείριση της ζώνης ευρώ κυρίως, αλλά τότε θα χρειαστεί ή θα μπορούσε να προβλεφθεί μια πολύ πιο θεμελιώδης αναθεώρηση της συνθήκης. Στο πλαίσιο αυτό, πού κινούνται συζητήσεις στο Συμβούλιο και σε σχέση με την τελευταία συμφωνία που έγινε για τον μόνιμο χαρακτήρα του μηχανισμού στήριξης. Αυτή νομίζω είναι η ερώτηση που θα σας υποβάλουμε και